Καλησπέρα, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Για γραφειοκρατικούς λόγους, ανεξάρτητους από τη θέλησή μας, δυστυχώς θα πρέπει μάλιστα να φύγω για τρία τέταρτα, ίσως τις πέντε και τέταρτο, ίσως πεντέμιση αν τα καταφέρω. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς που από τις πέντε και μετά θα είναι μαζί μας. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να φύγω για την Κινσάσα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η οθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Το πρόγραμμα ε, μοιράστηκε στις 23 Νοεμβρίου. Θα ξέρετε ότι σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες για την πρωτοβουλία των πολιτών. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Σήμερα όμως το απόγευμα ελπίζω να είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφος ε, Μέντες Δεβίγκου, ούτως ή άλλως και ο κύριος Νταφ ζητούν η Επιτροπή μας, πέρα από τα σημεία τα οποία έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη, να διενεργήσει και μια συζήτηση για τα συνταγματικά θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό. Εάν συμφωνεί η Επιτροπή, συμφωνείτε, δεν βλέπω αντιρρήσεις, θα μπορούσαμε να εντάξουμε και αυτό το σημείο και να το συζητήσουμε πριν από τις Ελπίζοντας πάντα να έχουμε και κάποιο χρόνο για να συζητήσουμε και τις τροπολογίες για την πρωτοβουλία των πολιτών, της έκθεσης για την πρωτοβουλία των πολιτών. Γιατί όπως σας είπα ήδη πριν, στις 5 θα ακούσουμε την παρέμβαση του Αντιπροέδρου και Επιτρόπου κ. Σεύκοβιτς για την ενεργοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας ε, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Συγγνώμη. Αύριο το πρωί πέρα από την ε, ψηφοφορία της έκθεσης Γκουρμάη Λαμασούρ, θα ψηφίσουμε και την έκθεση για τεμάκι για την ε, πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της, Ευρω... οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δύο εκθέσεις ε, του κυρίου Νταφ για την εκλογική διαδικασία και μια τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Όπως σας είπα, θα αναγκαστώ να φύγω πριν το τέλος της συνεδρίασης. Σας υπενθυμίζω ότι ήδη από τώρα, καλό θα ήταν αύριο να φτάσετε στη συνεδρίαση με, τα, με τις ηλεκτρονικές σας ε, κάρτες για την ψηφοφορία. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα τις χρειαστούμε ή όχι. Καλό είναι να μην χάσουμε χρόνο αν τις χρειαστούμε για να πάτε, να φύγετε, δηλαδή να τις βρείτε κτλ. Λοιπόν, αν συμφωνούμε με την ημερήσια διάταξη, περνάμε στον ανακοινώσει του Προέδρου. Ε, στις 9 Νοεμβρίου εγκρίθηκε η σύνθεση της ε, Επιτροπής μας που θα μεταβεί στην ε, Βουδαπέστη, της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας. Θα έχουμε άλλους δύο βουλευτές, την ε, κυρία Αλεξάνδρα Τέιν και τον Ζώσεφ Σάιερ, που είναι εκτός ποσόστοσης. Έτσι, ο κύριος Σάιερ που είναι Ούγγρος. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, μπορούμε να περάσουμε στο φάκελό σας. Εκεί θα δείτε ένα σημείωμα με κάποιες προκαταρτικές ημερομηνίε για τις συνεδριάσεις της επόμενης χρονιάς. Αποφασίσαμε για αυτές τις ημερομηνίε στη συνεδρίαση της 5ης ε, Οκτωβρίου. Πάμε στην έγκριση τώρα των ε, πρακτικών των ε, προηγούμενων συνεδριάσεων της 30 Σεπτεμβρίου, και τις 4 και 5 Οκτωβρίου. Ως ήθιστε, αν δεν έχετε παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Τώρα, με βάση τη μερίσια διάταξη που σας έστειλα, προβλέπετε η συζήτηση των τροπολογιών για την έκθεση Λαμασούρ και Γκουρμάη. Πριν από λίγο Είπαμε ότι συμφωνούμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Μπορεί να ξεκινήσει ο κύριος Μέντες Τεβίγκο για να συζητήσουμε τα θεσμικά θέματα και τα συνταγματικά θέματα, τις συνταγματικές πτυχές της ε, ε, διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού. Ο κύριος Μέντες Τεβίγκο. Νομίζω ότι όλοι μας περιμένουμε τη συζήτηση σε σχέση με την πρωτοβουλία των πολιτών. Νομίζω ότι είναι το κύριο αντικείμενο τη συνεδρίασή μα. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, μπορώ να παρεύω μετά, κύριε Πρόεδρο. Γιατί νομίζω το πιο σημαντικό θέμα στη συνεδρίασή μα αυτή τη βδομάδα είναι η αυριανή ψηφοφορία για την πρωτοβουλία πολιτών. Οι συγητέ έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καταλήξουν σε συμβαστικέ λύσει και εμεί ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να ακούσουμε τι προτάσει του. Σημαντικό είναι και το θέμα αυτό που αναφέρεται, αλλά θα ήθελα να το κάνουμε μετά από την πρωτοβουλία πολιτών. Γι' αυτό θα ήθελα η κυρία Γκουρμά και ο κύριος Λαμασούρ να μας παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να γίνει η συζήτηση αύριο και μετά μπορούμε να γυρίσουμε και στο θέμα του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Αυτά είχαμε πει και στην αρχή, είχα πει δηλαδή στην αρχή. Αλλά τελικά διάφορες φήμες με οδήγησαν στο να θεωρήσω ότι πρέπει να καθυστερήσουμε. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την έκθεση Γκουρμάη Λαμασού. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Ενημερωτικά σας λέω ότι έχουμε 60 τροπολογίες των συζητών. 144, ε, των ε, βουλευτών, 63 των, ε, ε, της Επιτροπής Αναφορών, 38 της Επιτροπής Πολιτισμού και 68 της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είναι άπειρες οι τροπολογίες καλό θα ήταν να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες, όπου μπορούμε, να περάσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Διάβασα τις τροπολογίες, πολλές είναι επανομοιότυπες. Ελπίζω λοιπόν οι συγητές μας να μας αναγγείλουν καλά νέα. Δηλαδή να μας πούν ότι μπορούμε να ε, υιοθετήσουμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. επίσης θα πρέπει να πάρουμε και μία απόφαση για τους διαπραγματευτές της Επιτροπής. Στις 13 ε, του μηνός, Δεκεμβρίου δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα για να πάει στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και τις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να κλείσει το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Και σε αυτή την Ολομέλεια θα πρέπει να αποφασίσουμε και τα της διαπραγμάτευσης. Τέσσερις βουλευτές είναι οι συγκητές μας, Wallace και Hefner, Ξέρετε ότι στο Λονδίνο και, το, και στο Μόναχο χιονίζει και άρα έχουν κλείσει τα αεροδρόμια και μπορεί να μην μπορέσουν να έρθουν από τις δύο αυτές πόλεις. Αλλά ε, ζητούν σε αυτή την ομάδα να συμμετάσχουν και όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων σε αυτή τη διαπραγματευτική ομάδα. μπορούν να μιλήσουν οι συγητές, τα, οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι των άλλων επιτροπών, ιδίως της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, που είναι παρόντες. Η κυρία Γκουρμάη θα μιλήσει πρώτη και συνεχεία ο κύριος Λαμασούρ. Ε, ή μάλλον όχι, ο κύριος Λαμασούρ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το παίξαμε στα ζάρια, εγώ θα κάνω την παρουσίαση και η κυρία Γκουρμάη θα βγάλει τα συμπεράσματα στο τέλος. Θέλω να σας υπενθυμίσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, την απαρχή αυτής της, στην απαρχή αυτής της συζήτησης ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία μιας ιδιαίτερα μακροσκελούς διαδικασίας. γιατί σε ό,τι αφορά τους εισηγητές της Συνταγματικής Επιτροπής και μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, έγιναν οι πρώτες εργασίες πριν από τις καλοκαίρινες διακοπές. Προτάσεις σας κύριε Πρόεδρε. Δημιουργήσαμε μία μονάδα κοινή συνεργασίας μαζί με τους δύο εισηγητές της Επιτροπής Αναφορών και ήταν η μέρη μας, οι επαφές οι οποίες τότε ήταν απλώς άτυπες μεταξύ μας με το, και με το Συμβούλιο καθώς και την Επιτροπή να λάβουν χώρα, να λαμβάνουν χώρα τακτικά ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες ήταν οι πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις και πού θα μπορούσαμε να σκοντάψουμε σε προσκόμματα. Αύριο μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, αν θέλει ο Θεός, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα έχουν πια αποκομίσει μια πολιτική εντολή ώστε να ξεκινήσει ο επίσημος τριγωνικός διάλογος τον οποίο έχουμε προβλέψει. Έχουμε προβλέψει συγκεκριμένα μια συνεδρίαση αύριο το απόγευμα, αμέσω μετά από την ψηφοφορία που θα γίνει το πρωί στην Επιτροπή μας και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην αρχή της επόμενης εβδομάδας ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε το πολιτικό χρονοδιάγραμμα όπως τονίσατε εσείς κύριε Πρόεδρε που έχει και συμβολική σημασία ώστε το Δεκέμβριο, ένα χρόνο μετά την θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, μετά από εργόδεις εργασίες, μετά από προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πράσινη Βίβλη και την συνεργασία όλων αυτών των φορέων να μπορέσουν οι δύο αρχές τα δύο σκέλη τη αρχή του προπολογισμού να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο με μία μονάχα ανάγνωση. Σε σχέση με τι αρχικέ προτάσει της Κομισιόν, η εργασία αυτή μα επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνίε ή να πλησιάσουμε ιδιαίτερα σε συμφωνίε που θα προσπαθήσουμε να τι μεταφράσουμε σε συγκεκριμένε τροπολογίες μαζί με την Τσίτα, ώστε για κάθε μία από τις τρεις φάσεις της διαδικασίας τις οποίες θα υπενθυμίσω τη φάση της κατα... κατάθεσης μιας πρωτοβουλίας, μετά τη φάση συλλογής των υπογραφών και της φάσης ε, κατά την οποία θα δίδεται συνέχεια σε μια πρωτοβουλία που έχει ήδη καρποφορήσει. Για την πρώτη φάση η μεγάλη καινοτομία που φέρουμε σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και σε σχέση επίσης με την πολιτική συμφωνία που είχε γίνει τον προηγούμενο Ιούνιο στο Συμβούλιο στο τέλος της Ισπανικής Προεδρίας. Η καινοτομία είναι ότι ουσιαστικά ε, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, απαρνούμεθα οποιαδήποτε προϋπόθεση σε σχέση με τον αριθμό πολιτών που θα πρέπει να υπογράψουν μία ε, πρωτοβουλία πολιτών για να μπορούμε να ελέγξουμε σε αυτή τη φάση το παραδεκτό αυτής της πρωτοβουλίας και έχουμε λοιπόν δύο χωριστές φάσεις. Η μία είναι η φάση της καταγραφής της πρωτοβουλίας και μετά η φάση του ελέγχου του παραδεκτού αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν ζητούμε λοιπόν να υπάρχουν 300.000 υπογραφές για να θεωρηθεί ότι μπορεί να καταγραφεί μία η πρωτοβουλία και να πάρει το δρόμο προς το 1 εκατομμύριο. Εφτά μονάχα φυσικά πρόσωπα, εάν υπογράψουν, μπορούν να συμπήξουν μια οργανωτική επιτροπή και φυσικά πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Ο αριθμός των 7 ε, συνδέεται με τον, αριθμό του, με τον ελάχιστο αριθμό χωρών από τις οποίες θα πρέπει να προέρχονται οι πολίτες που θα υπογράψουν αυτήν την πρωτοβουλία. Το κατόφλι αυτό, το οποίο για την Κομισιόν και το Συμβούλιο έπρεπε να είναι το 1 τρίτο των κρατών μελών, εμείς θέλαμε να είναι το 1 πέμπτο η τελική απόφαση θα είναι μάλλον ένα τέταρτο, αλλά ο στόχο είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό πολιτών που αντιστοιχεί στον αριθμό των ελάχιστων των κρατών μελών. Είτε είναι 6, είτε είναι 10, είτε είναι 12, είτε είναι 5. Θα πρέπει να είναι άνθρωποι. Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, δεν μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα. Γιατί δεν είναι τέτοιο το πνεύμα της συνθήκης, ούτε και το γράμμα της συνθήκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νομικοί φορείς δεν μπορούν να ενθαρρύνουν, να πατρονάρουν, να παρακινήσουν, να χρηματοδοτήσουν ή ακόμα και να αντιταχθούν σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Αλλά τα πραγματικά τα φυσικά άτομα θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτή την πρωτοβουλία μέσα από τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών, μάλιστα <clears throat> για να είμαστε πιο σαφείς, το γιατί χρειάζεται να καλύπτουν μια ελάχιστη ηλικία. Από όλους αυτούς, από τους κοινοβουλευτικούς, από τους... Ε, μάλλον από αυτούς εκτός των κοινοβουλευτικών, των εθνικών και των ευρωπαίων, μπορεί να προέλθει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θέλουμε να είναι στο δυνατόν πιο απλή αυτή η διαδικασία, στα μέτρα του δυνατού. Αναφέρθηκα λοιπόν <clears throat> τον αριθμό των ελάχιστων των κρατών που θα πρέπει να τηρείται και θέλω να προσθέσω σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση, δηλαδή την κατάθεση της πρωτοβουλία πολιτών. Να σας κάνω μερικέ ε, διευκρινήσεις που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές για την πρόταση αυτή. Πρώτα απ' όλα, προσκαλούμε καταρχήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα τεχνικής αρρωγής για τους συντάκτες πρωτοβουλειών πολιτών υπό τη μορφή ενός γραφείου υποδοχής ή αγγλιστή help desk. Διότι αναγνωρίσουμε ότι αν θέλουμε αυτή η διαδικασία πράγματι να είναι πρόσφορος και να χρησιμοποιείται από τους πολίτες οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι σε κάποιον συγκεκριμένο φορέα, δηλαδή δεν ανήκουν σε συνδικάτα, πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κτλ. Η ιδέα αυτή αφορούσε κυρίως τους πολίτες οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι λοιπόν, η ενέργεια της πρωτοβουλίας πολιτών, θα πρέπει να έχουν μια διοικητικοτεχνική αρρωγή και ως, αντιστά, ως αντίτιμον κατά κάποιο τρόπο αυτού του δικαιώματος να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το γραφείο αρρωγής, θα φέρουν και την απόλυτη υποχρέωση διαφάνειας. σε ό,τι αφορά την οικονομική και πολιτική τους υποστήριξη. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιοδήποτε λόμπι, οποιαδήποτε εκκλησία, πολιτικό κόμμα μπορούν να ενθαρρύνουν οικονομικά, μέσω των μέσων ενημέρωσης, χρηματοδοτικά μια πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει οι πολίτες οι οποίοι υπογράφουν αυτή την πρωτοβουλία να ξέρουν ακριβώς ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και ποιος την υποστηρίζει. Απόλυτη διαφάνεια λοιπόν φιλική προς τους πολίτες και διάφανη πρέπει να είναι η πρωτοβουλία. Και φιλική προς τους υπογράφοντες. Δεν πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να τύχει κατά χρήσεων. Και έρχεται η φάση της, της συλλογής των υπογραφών. Ποιος μπορεί να υπογράψει. Η πρότασή μας είναι ότι Πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Εδώ μα δεσμεύει η συνδίκη τη Λισαβόνα. Δεν μπορούν να υπογράψουν πολίτε τρίτων χωρών. Θέσαμε το ερώτημα της ελάχιστης ηλικία. Εμείς προτείνουμε μια κοινή λύση για όλα τα 16 ετών. Αλλά δεν πρέπει να αυταπατώμεθα. Αυτή η λύση, ακόμα κι αν γίνει δεκτή από εμά δεν θα γίνει δεκτή από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία, θα μα το επιβεβαιώσει και ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου αν θέλετε. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο που θεωρούν ότι η αντίστοιχη ηλικία θα πρέπει να είναι η ηλικία που δίδει το δικαίωμα του εκλέγην και η οποία καθορίζεται από το εκλογικό δίκαιο και σε 26 χώρες η ηλικία αυτή είναι στα 18 και μόνο στην Αυστρία από τους 16 άνδες. Και άνω. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και δεν πρέπει να τρέχουμε πολλές ψευδεστήσεις σε σχέση με την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Προσθέσαμε και την ιδέα ότι η Κομισιόν θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των οργανωτών των πρωτοβουλίων πολιτών ένα ε, ελεύθερο λογισμικό λογισμικό ανοιχτή πηγή, όπω λέγεται, για να, μπορεί, να μπορούν να συλλέγουν υπογραφέ. Και φυσικά τώρα έχουμε ένα μεγάλο, έχουμε το μόνο πραγματικό πολιτικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτό είναι η επαλήθευση των συλλεχθισών υπογραφών και οι απαιτήσει ορισμένων κρατών μελών σε σχέση με τον έλεγχο της ταυτότητας των υπογραφώντων για να αποφύγουμε ε, υπογραφές οι οποίες είναι πλασματικές ή οι οποίες είναι διπλές. Το ίδιο άτομο υπογράφει δύο φορές. Για πρακτικούς λόγους. Ο έλεγχος των υπογραφών δεν μπορεί να γίνει από τις εθνικές διοικήσεις στα κράτη-μέλη με την δική τους ευθύνη και επίσης στα κρατημέλια έχουμε διαφορετικές παραδόσεις αλλά και διαφορετικές, αρκετά διαφορετικές νομικές βάσεις για τον έλεγχο της ταυτότητας των υπογραφώντων. Όπως γίνεται παραδείγματος χάρη όταν πηγαίνει κανείς στην κάλπη για να ψηφίσει. Έχουμε λοιπόν προτείνει μια συμβαστική λύση στον τελευταίο άτυπο τριγωνικό διάλογο. Κάνουμε αυτή την πρόταση προς το Συμβούλιο που θα την εξετάσει νομίζω σήμερα το πρωί το πράτη ήδη. Αλλά είναι απαραίτητο και οι δύο πλευρές να δείξουμε αμοιβαία κατανόηση γιατί τα σημεία εκκίνησης ήταν πολύ απομεμακρυσμένα. Από την, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε η αίτηση να υπάρχει ταυτόσιμος έλεγχος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες για τον έλεγχο της ταυτότητας των υπογραφώντων και το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τυπικών διαδικασιών. Από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ε, δυνατότητες ελέγχου από κάθε χώρα, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες φυσικά οι οποίες θέλησαν να υπάρξει ένας πιο αυστηρός έλεγχος ταυτότητας. Για την τρίτη φάση τώρα, δηλαδή. Ποια θα είναι η συνέχεια η οποία θα μπορούσε να δοθεί σε μια πρωτοβουλία η οποία έχει συλλέξει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Εδώ ερχόμαστε στην ε, αρχή της βασικής ευθύνης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει το μονοπόλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Επομένως, αυτή είναι ο φορέας ο οποίος εξασφαλίζει το σεβασμό του συνόλου των συνθηκών επομένω και των συγκεκριμένων άρθρων που θεσπίζουν την πρωτοβουλία πολιτών. Η Κομισιόν λοιπόν έχει την ευθύνη να αποφασίσει και να δώσει μια νομοθετική ενσάρκωση ή όχι στην πρόταση η οποία έρχεται από την πρωτοβουλία πολιτών. Αλλά προβλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει η Κομισιόν να απαντήσει στην πρωτοβουλία μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο και δεύτερον να προβλέπει ο κανονισμός αυτός ένα δικαίωμα των πολιτών των οποίων έχει ευδοκιμήσει η πρωτοβουλία τους να υπάρξει και δημόσια ακρόαση σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή. Με λεπτομέρειες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί γιατί θα πρέπει να τις συζητήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ποιος οργανώνει την ε, ακρόαση, αν το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το κάνει το Κοινοβούλιο. Εάν μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιοι κοινωνικοί φορείς, κοινωτικοί φορείς όπως είναι η, περιοχή, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο διαμεσολαβητής παραδείγματος χάρη πέραν των βασικών θεσμών μπορούν να συμμετάσχουν. Όλα αυτά βέβαια είναι μια σημαντική καινοτομία με στόχο να εξασφαλίσουμε για όλους τους οργανιτές πρωτοβουλειών οι οποίες έχουν ευδοκιμήσει ότι τουλάχιστον θα ακολουθήσει μια δημόσια συζήτηση για την πρότασή τους, ότι θα έχουν το δικαίωμα τη δημόσια συζήτηση για την πρότασή τους και φυσικά υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τέλος και το ίστατο σημείο, ξέρω ότι αυτό είναι ένα σημείο για το οποίο εσείς κύριε Πρόεδρε είχατε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να καθορίσουμε ένα χρονικό ορίζοντα, μια προθεσμία για την θέση σε εφαρμογή αυτού του κανονισμού, γνωρίζουν ότι ο κανονισμός αυτός, αν εγκριθεί το Δεκέμβριο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου, γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν και εφαρμοστικές διατάξεις για ό,τι αφορά το, τη φάση 2 της διαδικασίας, δηλαδή τη συλλογή των υπογραφών. Φυσικά επιθυμούμε το ταχύτερο δυνατό οι πολίτες να έχουν αυτό το σύστημα στη διάθεσή τους, αλλά τίθεται το ερώτημα πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για την εφαρμογή αυτού του συστήματος, της πρωτοβουλίας των πολιτών και επίσης, εφόσον το επιθυμούμε, μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προβούμε σε μία επισκόπηση και αναθεώρηση του συνόλου αυτής της διαδικασίας, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα που θα έχουμε αντλήσει από την πρώτη φάση εφαρμογής της διαδικασίας αυτής. Είναι πολύ πιθανό ότι κάποιες από τις διατάξεις τις οποίες προβλέπουμε τώρα θα φανούν ότι δεν είναι πάρα πολύ λειτουργικές, ότι δεν είναι προσαρμοσμένες προς την πραγματικότητα, ότι θα χρειάζονται βελτίωση, ίσως λοιπόν σε τρία, σε 5 χρόνια υπάρχουν διαφορετικές τροπολογίες, θα πρέπει να προβούμε σε μια επισκόπηση. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε τα κύρια σημεία στα οποία καταλήξαμε μετά από την ενδελεχή αυτή εργασία και είμαι σίγουρο ότι οι τροπολογίε οι οποίε θα τύχουν καταθέσεω από του συναδέλφου έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν έτσι περισσότερο το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρο. <clears throat> Ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ ευφυή, πάρα πολύ σημαντική εργασία του κυρίου Λαμασούρ και τη κυρία Γκουρμάη, στην οποία τελευταία δίδω τώρα τον λόγο. Thank Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε opportunity Να uh, uh, uh, το συζητήσουμε ναι πριν γίνει αύριο η ψηφοφορία για να δούμε και να διαπιστώσουμε πόσο έχει κινητοποιήσει του συναδέλφου η ανάγνωση αυτού του κειμένου. Έχουμε συγκεντρώσει μια πολύ πλατιά συνένεση, αλλά και η σημερινή συνεδρίαση θα μας καθοδηγήσει περαιτέρω. Δυστυχώ οι συνεισηγητέ μας δεν είναι εδώ, Ζωάρη και Νταϊάννα, για να τα συζητήσουμε. Όμως ευτυχώ και ο Πρόεδρος και η Ομιλούσα κάναμε όλοι προ το χέρι μας για να μπορέσουμε μέσω Φραγκφούρτη να έρθουμε εδώ και που πιστεύαμε ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Βεβαίω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουμε πάρα πολλέ τροπολογίε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν κινητοποιηθεί όχι μόνο στην ε, θεσμική επιτροπή μας, αλλά και στις άλλες επιτροπές. Είμαστε του δύο κύματος και το ότι έχουμε τόσο παρομοιάζουσες τροπολογίες δείχνει όλη αυτή η διαδικασία πόσο καλά και ο Αλέν και ο Μιλούσα και άλλοι δύο συνεισηγητές ελπίζουμε ότι θα τα βρούμε και θα επινοήσουμε κάποιες συμβαστικές πλήρες τροπολογίες. Τώρα έγινε αυτή η πλήρης ε, εισήγηση για, για την όλη διαδρομή και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά το οποίο δείχνει ότι αυτή η καινούργια ευρωπαϊκή επινόηση πρόκειται να μας βοηθήσει στην συμμετοχή δημοκρατία. Θεωρήσαμε ότι έχουμε ευθύνη να καταλήξουμε σε κάτι το αξιόπιστο για τον Ευρωπαίο. Οπότε περιμένω και από εσάς ιδέες για να πάμε παραπέρα. Βεβαίω και με τους ηγητές προσπαθούμε να κλείσουμε κάποιες ε, συμβαστικές προπολογίες αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή η έκθεση θα είναι μια ευκαιρία να κλείσει το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Ήδη έγινε άτυπη συνάντηση με Κομισιόν και Συμβούλιο. Οπότε με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τη Συμβουλική Επιτροπή για την τόσο αγαστή συνεργασία, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ε, Βέβαιως και όλοι υπεύθυνα παίρνουμε αποφάσεις, οπότε θα αποδειχθεί από τη δουλειά μας ότι η Επιτροπή μας είναι ικανή να επιτελεί πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά να σε ευχαριστούμε και εσένα και τους άλλους αδέλφους που βοηθήσατε για αυτό το τόσο αξιόλογο έγγραφο. Να είναι όσο γίνεται πιο δυναμικό, πιο αναβαθμισμένο με τις τροπολογίες σας και αυτό αφορά και την Επιτροπή μας. Οπότε και όταν έρθει η ώρα σύντομα να έχουμε την επέτειο της νίκης της Λισαβόνας, τότε θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Πρώτος θέλει να μιλήσει. Η συνάδελφος Τούν από την Επιτροπή Πολιτισμού. Μπορώ να μιλήσω. Α, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, δεν έχουμε μετάφραση. Δεν έχουμε δερμηνία. Έχουμε αλλά δεν το είδε η ομιλήτρια. Οπότε θέλω να σας πω ότι από κοντά παρακολούθησε τις εξελίξεις και συνέταξα μία γνωμοδότηση για την Επιτροπή των Πολιτιστικών Ζητημάτων και ίσως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε μια που η τροπολογία αυτή προέρχεται από συναδέλφους από την ίδια πολιτική ομάδα. Μιλάμε για 119, μιλάμε για αυτή την τροπολογία της Πολιτικής Επιτροπής η οποία πάει λίγο παραπέρα και είναι το 119 επαναβαλλοντήτρια στο κείμενο το οποίο έχετε που αναφέρεται σε αυτή την Επιτροπή των Πολιτών όπως προαναφέρθηκε από κάποιον προηγουμένως έχω εδώ το πολωνικό κείμενο και εσείς έχετε το κείμενο στη γλώσσα σας Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι σημαντικό εάν θέλουμε. Σε αυτό το μέσο άσκηση πολιτικής να το προσδώσουμε με ένα φιλικό στον πολιτή χαρακτήρα και να διαπνέεται αυτό το χαρακτήρα του Κοινοβουλίου ως άμεσα εκλεγμένο οργάνο γιατί κάποιοι συνάδελφοι εδώ με τους οποίους το κουβεντιάσαμε είπαν ότι εάν βγουν από το παιχνίδι οι βουλευτές τότε θα έχουμε πολίτες α και β κατηγορίας. Άρα να συμπεριφθούμε και εμείς, μια που ήδη έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα για να νομοθετούμε. Ο επομένως έτσι θα καλυφθεί και αυτή η περίπτωση που αποσκοπούσε σε αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα να έχουν την πλατφόρμα την νομοπαρασκευαστική και γι' αυτό θα πρέπει η Οργανωτική Επιτροπή να μην συμπεριλαμβάνει βουλευτάς. Για φανταστείτε, κάποιοι από εμά δεν καταφέρουμε ό,τι θέλουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε με παρακαμπτήρια εδώ τέλο πάντων θέλουμε να περάσουμε αυτό το οποίο θέλουμε με την πρωτοβουλία των πολιτών. Επόμενο λόγο, ο απόλυτο λόγο είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για τα νομοθετήματα, οπότε και ταυτόχρονα προτείνει κάτι άλλο η Επιτροπή των Πολιτών. Δηλαδή προτείνει ένα νομοθέτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί. Επομένω, θα έχουμε του ίδιου οι οποίοι θα ζυγίζουν και θα αξιολογούν, οι οποίοι ταυτόχρονα θα είναι και στην Οργανωτική Επιτροπή. Καταλάβετε τι λέω. Όχι, ναι, ναι. Λέει ο κ. Μέντε Δεβίγκο, νεύοντα καταφατικά. Α, δεν κατάλαβα, δεν, δεν ξέρω αν σα τα λέω αρκετά. Ξεκάθαρα. Ωραία, ευχαριστώ. Και ο τελευταίος λόγος, το τελευταίο επιχείρημα με το οποίο θέλω να σας πείσω σχετικά με την τροπολογία μου είναι ότι θα ήταν πολύ αξιόλογο το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους. Είναι και τόσο αξιόλογη αυτή η πρόταση για τη συνθήκη της Λισαβόνα. που θα πάει χαμένη. Άρα στο χέρι σας είναι να την εκμεταλλευτείτε και οι άλλοι επίσης. Να αξιοποιήσουν τους στόχους της συνθήκης και αυτό επίσης είναι ένα μέσο προς χάρη του πολίτη και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει σωστή χρήση του. Δεν είναι κάτι το οποίο το, το, το, το, φτιάξαμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα ολίγα για να σας πείσω σχετικά με την τροπολογία την οποία κατέβασα στην Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και η οποία πάει λίγο παραπέρα από την ήδη προταθήσα 119 των συναδέλφων αυτή τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος Ντάφ. Καλησπέρα Πρόεδρε, καλησπέρα και όλους και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να κλείσει το θέμα ή δυνατόν σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά δεύτερον να μην γίνει εις βάρος της ποιότητας του νομοθετήματος ή της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας γιατί υπάρχουν κάποια θέματα ουσιαστικά τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Πέντε σημεία θέλω να σας αναφέρω. Πρώτον, άρθρο 2, παραγράφος 2. Εκεί αντιμετωπίζεται το ζήτημα του τι είναι προσυπογράφουν το ψήφισμα ή τέλο πάντων το κείμενο της πρωτοβουλίας. Δεν θέλουμε να υπάρχει δυσμενή διάκριση και να διώγνουμε ή να εξαιρούμε, να αφήνουμε απ' έξω κάποιους οι οποίοι νόμιμα διαβιούν και κατοικούν στην επικράτεια της Ένωσης. χωρίς να έχουν την ηθαγένεια κάποιου κράτους μέλους. και οι οποίοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν στους του νόμους και να καταβάλουν φόρους. Κράτη μέλη της μας. Οι οποίοι ενδιαφέρονται να υπάρχει κοινωνική ευημερία οπότε. Έτσι, μπορούμε να καλύψουν και κάποιους που έχουν το δικαίωμα του εκλέγην κατά τις ευρωεκλογές, διότι το εκλογικό σώμα για τις ευρωεκλογές δεν έχει μόνο πρόσωπα που, είναι, που έχουν την ηθαγένεια κρατών μελών, αλλά και εκείνους οι οποίοι προβλέπεται ότι μπορούν να εγγραφούν σε εκλογικούς κατάλογους για τις σχετικές εκλογές. Χωρίς βέβαια αυτό να ισχύει με μέρος τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα υπάρχει άλλη μια δεύτερη και μάλλον ευρύτερη κατηγορία προσώπων που αφορούν ε, φερειπίν την περίπτωση των, των μελών της ρωσικής μειονότητας της Λετωνίας. 20% του πληθυσμού. Επίσης τους Τουρκοκυπρίους και άλλους που σήμερα με την εθνική νομοθεσία δεν προβλέπεται η συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθε της Ένωση. Και άρα εμείς εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιλάβουμε όσο γίνεται περισσότερους. Επομένω, να δούμε κατά πόσο γίνεται μια διάκριση εδώ μεταξύ αυτών που απολάβουν το προνομίο του να έχουν την ηθαγένεια κάποιου κρατούς μέλους. Και από την άλλη μεριά, εκείνων οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλους χωρίς να έχουν την ηθαγένεια και για αυτό υπέβαλα την τροπολογία 111. Σε σχέση με τη διατύπωση ορισμού του οποίου μπορεί να προσυπογράψει το κείμενο της πρωτοβουλίας και ε, επιδιώκω να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή αυτού του άρθρου του ορισμού. Επίσης, άλλο, που ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι κάτι το οποίο αφορά το πεδίο εφαρμογή στο βελληνικές της πρωτοβουλίας των πολιτών σε σχέση με το άρθρο 4 παράγραφος 3. Εκεί όπου οι συνεισηγητές θέλουν να δώσουν ένα, μια νέα ερμηνεία στη σχετική ρήτρα της συνθήκης, σχετική διάταξη συνθήκης, αλλά αυτή η ερμηνεία να είναι πιο στενή. Ορίζει η συνθήκη ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες ευρύτατος ορισμός και μεταξύ άλλων καλύπτεται και η αρμοδιότητα τροποποίησης των συνθήκων. Επίσης ορίζεται κατά δεύτερο λόγο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα στη διακριτική ευχαίρεια να απόκειται το να μπορεί να δώσει συνέχεια σε, αυτή την, σε αυτό το αίτημα των πολιτών σε σχέση με κάποια εφαρμοστική των συνθηκών πράξη, αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό θα ήταν το σχέδιο οδηγίας ή σχέδιο κανονισμού. Κάποια νομοθετική πρόταση. Τέλος πάντων. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε και θα έπρεπε να δοθεί μια άλλη ερμηνεία. Νομίζω αυτή την οποία πεδίωκαν οι συντάκτες της συνθήκης. Δηλαδή να καλύπτεται και η πρόταση τροποποίησης της ίδιας συνθήκης. Σαν αναθεωρησή της και από ό,τι υποψιάζομαι πρωτοβουλία των πολιτών θα μπορούσε να απευθύνεται προς εμάς και να ζητεί αναθεώρηση της συνθήκης. Και είναι πολύ αρνητικό. Αποστερεί από κάθε νόημα την πρωτοβουλία το να μην αποδεχθούμε μια τέτοια πρωτοβουλία με τέτοιο περιεχόμενο. Τρίτον, το τρίτο θέμα αφορά γιατί θεωρούμε φθήνους αναλογικότητας. Όσον αφορά κάποιους που θα πρέπει να μπορούν να υπογράψουν πρωτοβουλία που ξεκινά σε άλλο κράτος μέλος και έχω την τροπολογία 76 όπου λέω ότι θα πρέπει να δοθεί ένας στεγανός ορισμός. Και σας παραπέμπω στη συμβαστική τροπολογία 1, 0-1 τέλος πάντων, αλλά και στις τροποποίησεις του σχεδίου κειμένου όπως τις πρότειναν οι συνεισηγητές. Τέταρτον, αυτό το θέμα της συνέχισης της πρωτοβουλίας, συνέχιση μπορεί να έχει μια πρωτοβουλία, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει μία δημόσια ακρόαση. Σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι αναγκαίο, σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι επιθυμητό. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σουρεαλιστικό. Θα είναι σπατάλη χρόνου και χρήματος. Θα πρέπει εδώ να αφήσουμε το περιθώριο της διακριτικής ευχαίρεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να επιλέγει εκείνη για το κατά πόσον θα οργανώνει μια τέτοια δημοσία κρόση ή ου. Τελευταίο. Αφορά την τροπολογία της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ε, επί της 31ης παραγράφου. Προτείνεται να επικουρείται η Επιτροπή από μία άλλη Επιτροπή που να έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε με αυτό το ανεξάρτητο εδώ σε αυτό το σημείο. χωρίς να ψεύγουμε τώρα στις λεπτομέρειες, να μην υπερβάλλουμε και κάνουμε μια περίπλοκη ρύθμιση χωρίς να χρειάζεται γιατί είναι σχετικά απλό το να πούμε σε ποιες περιπτώσεις ε, επιβάλλεται να γίνει ή ου μια δημόσια πρόβαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Ο κύριος Γκουερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, την πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα της πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή μας, ο πρόεδρος μας ο κύριος Κασίνη, έκανε μια σκέψη και τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία για να προωθήσει την έννοια του Ευρωπαίου ηθαγενούς, του Ευρωπαίου πολίτη για να μπορέσουν να έχουν οι πολίτες, τα φυσικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους και ότι αυτό δεν ήταν καθαρά και μόνο ένα θεσμικό και διακρατικό εγχείρημα, ένα εγχείρημα μεταξύ πολιτικών εξουσιών, αλλά και κάτι το οποίο είχε άμεση επίπτωση για, την, ε, για τους απλούς πολίτες και τους έδινε την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. είναι μία από τις ευτυχείς στιγμές που καμιά φορά έρχεται και γίνεται πραγματικότητα. Αν αύριο ψηφίσουμε και εγκρίνουμε την εντολή των εισηγητών για να διαπραγματευτούν για τα θέματα αυτά, τότε θα το κάνουμε ακριβώς ένα χρόνο μετά από την θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και θα επιτρέψουμε να υπάρχει μια θεσμική εξέλιξη μετά από την θέση εφαρμογή τη Συνθήκη Λισαβόνα, η οποία θα συνοδεύεται από μια ενίσχυση τη δυνατότητα των πολιτών να υποστηρίξουν αυτή τη θεσμική εξέλιξη. Και στρέφομαι σε κάτι που είπε ο κύριος Νταφ. Όταν μιλάμε για πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να διατρέχει την έννοια του πολίτη η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται από Ευρωπαίους πολίτες, από πολίτες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να ενδιαφέρει, μπορεί να ωφελεί και θα ωφελεί όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι οποίοι δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Επομένως, μπορεί ο Ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει το δικαίωμά του σε οποιοδήποτε κράτος στο, του χώρου αυτού στο οποίο είναι Ευρωπαίος πολίτης. Εγώ εκεί που συμφωνώ με τον κύριο Νταφ είναι ότι δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα της πρωτοβουλία πολιτών στο βωμό της ταχείας έγκρισης αυτού του κανονισμού. Νομίζω όμως ότι έχουν οριμάσει αρκετά τα πράγματα, έχει υπάρξει πλήρη συζήτηση στην Επιτροπή μας, η συζήτηση που προετοίμασαν οι εισηγητές και έχουμε τη δυνατότητα στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν στον μελλοντικό τρίλογο να βοηθήσουμε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η πρόταση. Επομένως αυτό το οποίο εξακολουθεί να είναι ασαφές αυτή τη στιγμή δεν είναι επειδή είναι ασαφές από την φύση του. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών θέσεων θα πρέπει να υπάρξει κάποια επίλυση. Και νομίζω ότι η στιγμή να το κάνουμε αυτό είναι αύριο στα πλαίσια της ψηφοφορίας που θα γίνει για αυτή την πρωτοβουλία πολιτών. Αν δεν έχουμε λοιπόν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα ακόμα, δεν επειδή πλανάται ακόμα μια ασάφεια, αλλά επειδή έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, οι οποίες μπορούν να επιληθούν μονάχα με μια διαδικασία ψήφισης. Πιστεύω πάντως ότι πρέπει να δώσουμε και κάποια ευελιξία στους εισαγητές, ώστε να μπορέσουν να διαπραγματευτούν με πλήρες εξουσίες μετά από την έγκριση αυτής της, ε, της πρότασης για την πρωτοβουλία πολιτών. Και γι' αυτό ξαναγυρίζω σε κάτι που ανέφερε ο πρόεδρος μας. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, αλλά ουσιαστικά τρία ή τέσσερα επίμαχα θέματα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε και γύρω από τα οποία περιστρέφεται η πλειοψηφία των τροπολογιών. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν αν κάποια πολιτική ομάδα έχει κόκκινες γραμμές για κάποια από αυτά τα θέματα να το εκφράσει αυτό, να το κάνει σαφές και στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πιστεύω θα είναι δύσκολο να γίνει δεκτή ως ελάχιστη ηλικία σε όλη την Ευρώπη η ελάχιστη ηλικία των 16 ετών αλλά σαν διαπραγματευτικό όπλο μπορεί να είναι πράγματι πάρα πολύ χρήσιμο για να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτή τη πρωτοβουλία. Ο κ. Λαμασούρ επίση αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει και αυτό στις ακροάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν. Βέβαια πρέπει να πούμε πώς, με ποιο τρόπο. να συμμετέχει με το να οργανώσει ακροάσεις αυτές στο Κοινοβούλιο με την παρουσία της Κομισιόν, να συμμετέχουν μέλη της Συνταγματικής Επιτροπής σε αυτές τις ακροάσεις. Τι από όλα αυτά. Και τέλος, για, το... για την προθεσμία εφαρμογής στην πράξη αυτή του κανονισμού. Νομίζω ότι θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι χρειαστήκα μόνο ένα χρόνο για να θέσουμε στην εφαρμογή αυτή την πρωτοβουλία. Αν, καθα... αν καθυστερήσουμε πολύ την ε, υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, θα θεωρήσουν πολύ ότι <clears throat> αντιμετωπίζουμε πολύ πιο γρήγορα άλλα θέματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν τόσο τους πολίτες και καθυστερούμε αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες. Αν λοιπόν καθορίσουμε μια προθεσμία, έξι μήνες που έχω όπως είπαν οι για τα κράτη-μέλη, για να κάνουν όλες τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή αυτής της ε, ρύθμισης, νομίζω ότι θα είναι επαρκής χρόνος και δεν χρειάζεται να παρατείνουμε περαιτέρω αυτή την προθεσμία. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ε, χρονική προθεσμία που αναφέρουν οι συγητές για την αναθεώρηση των ρυθμίσεων και τρία χρόνια μου φαίνεται καλύτερη προθεσμία από τα πέντε χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια συσσωρευμένη κατά κάποιο τρόπο θέληση για να εφαρμοστούν οι διαδικασίες αυτές της πρωτοβουλίας πολιτών. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες λοιπόν θα διατυπωθούν ήδη από την αρχή της διαδικασίας και μετά από τρία χρόνια θα έχουμε αρκετή πληροφορία για να καταλάβουμε πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Μετά από την παρέμβασή σας, μια και αναφερθήκατε σε κάποιες προηγούμενες ε, παρατηρήσεις που έκανα εγώ, θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι το πρόβλημα της ηλικία θα πρέπει να επιληθεί. Μπορούμε βέβαια να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν για την ελάχιστη ηλικία ή να πούμε ότι θα ισχύει η ηλικία για όλους των 18 ετών. Τώρα, για τη διαφορά ανάμεσα στα 16 και στα 18 χρόνια. Σε ορισμένες, ε, σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχει δυνατότητα να εκλέξει κανείς, ε, να ψηφίσει μάλλον κανείς ε, στο ένα σώμα της Βουλής στα 16 και, στο, και σε κάποιο άλλο, στο άνω σώμα ας πούμε, ε, στα 18. Το θέμα της Ευρώπης δεν είναι θέμα φεδρό, δεν είναι θέμα αστείο. Χρειάζεται ίσως μια μεγαλύτερη ε, οριμότητα. Ίσως καλύτερα λοιπόν 18 χρονών να είναι ο πολίτης που ψηφίζει ή που υπογράφει, εν πάση περιπτώσει, από 16. Και για το θέμα της ηθαγένειας, συμφωνώ με τον κύριο Γκερέρο. Η πρωτοβουλία θέλει να υπογραμμίσει την ιδιαίτερη σημασία της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Για να μην χαθεί λοιπόν αυτό το στοιχείο, ε, ίσως δεν μπορούμε να δώσουμε, να ανοίξουμε αυτή την πρωτοβουλία σε όλους τους πολίτες αρκεί να διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης για την προθεσμία να κάνω κάποια παρατήρηση. Υπάρχουν κάποιες χώρες μεταξύ των 27 που δεν έχουν κανένα μηχανισμό ε, άμεσης συμμετοχής. Εμείς, ας πούμε, στη χώρα μου έχουμε το δημοψήφισμα. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια καινοφανή στοιχεία στον τρόπο που θα παρέμβουμε ως πολίτες. Στην Ιταλία, ας πούμε, προβλέπεται ότι καμία, κανένα αδίκημα δεν μπορεί να τιμωρηθεί αν δεν υπάρχει αναλογική ποινή για αυτό το αδίκημα. Δίκαιη και αναλογική ποινή. Στο σημείο 13 της πρότασής σας λέτε ότι οι οργανωτές, οι οργανωτές της πρωτοβουλίας, λέτε στην αρχή αρχή, είναι υπεύθυνοι ε, και έχουν και αστική ή ποινική ε, ευθύνη για ψευδείς δηλώσεις και υπογραφές. Παραπέμπουμε λοιπόν στον ποινικό ε, κώδικα. Νομίζω ότι οι σημερινοί ποινικοί κανόνες που υπάρχουν δεν μας καλύπτουν. Υπάρχει και ένας άλλος παραλογισμός. Η Κομισιόν με βάση την πρόταση, έχει 6 με 9 μήνες για να εκπονήσει ένα σύστημα ε, ηλεκτρονικής καταχώρησης. Ενώ τα κράτη έχουν μόνο 6 μήνες, κάτω από, δηλαδή λιγότερο από τους 9 μήνες, για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή αυτής της απόφασης για τη λειτουργία του Ινστιτούτου στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Τα πράγματα είναι σημαντικά. Αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών καλό θα ήταν να, να τη διευκολύνουμε για να την ε, δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες οι πολίτες μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολεμικές Θα πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε πού είναι οι διαφωνίες. Επίσης, για αυτό το Ινστιτούτο που προτείνεται, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα, όλα τα θέματα που το αφορούν ήδη από την αρχή, για να μην δημιουργηθούν και γι' αυτό πολεμικέ περτέ. Ε, τα κάνω όλα αυτά τα σχόλια, γιατί αύριο δεν θα είμαι. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόμπς. Ευχαριστώ. Δεν είναι παραδεκτή μια πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει να χτίζεται από καταχρηστικότητα ή έλλειψη σοβαρότητα ή να αντιβαίνει κατάφορα τη Ευρωπαϊκή αξίες. Τα είπαμε εδώ και άλλη φορά. Αυτό είναι ο στόχος και από την άλλη μεριά θέλουμε να είναι ελεύθερο ο προβληματισμό και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίση, σε σχέση με τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού τη ίδια, προτείνεται ότι εάν δεν υπάρξει σοβαρότητα ή ε, καταγραστική χρήση ή αντίθεση στι αξίε, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί όταν κατατίθεται και πρωτοκολλείται άρθρο 2 παραγωγή 4 που λέει ότι η πρωτοκόλληση θα πρέπει να γίνεται αμελητή πλην εάν και παραπέμπει στην παραθέτρια και 4 σε, ακριβώς σε αυτά τα ελαττώματα του κειμένου. Επίσης, στο δεύτερο παράρτημα ορίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια νομική βάση την ώρα τη πρωτοκόλληση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα γίνει πρωτοκόλληση αν θεωρεί η Επιτροπή ότι δεν υπάρχει νομική βάση. Άρθρο 8. Εκεί ορίζεται ότι η απόφαση επί του παραδεκτού θα λαμβάνεται μόλις έχουν προσυπογράψει 300. Τι γίνεται με αυτό, αυτό συνάδει προς το υπόλοιπο που είπαμε, δεν το είχα προσέξει προηγουμένως. Μέντες Κύριος Μέντες κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το θέμα το οποίο μας ε, συγκεντρώνει εδώ σήμερα και η αυριανή ψηφοφορία θα έχουν μια τεράστια σημασία πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν πολλές προσδοκίες σε σχέση με το ζήτημα αυτό και το αξίζει το θέμα αυτό και δεύτερον γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς τους ίδιους πάρα πολύ αυτό το θέμα. Θυμάστε όλοι την ε, συντακτική συνέλευση η οποία κατέστη πραγματικότητα χάρη στην κοινή δράση εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών. Καταφέραμε την τελευταία στιγμή να εγκριθεί στο σχέδιο της συνταγματικής συνθήκης η έννοια της πρωτοβουλίας πολιτών. Από εμά έχει ξεκινήσει λοιπόν και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όπως είπαν και πολλοί άλλοι που καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο από την ε, θέση εφαρμογή της συνδίκη Λισαβόνα να βρεθούμε σε αυτό το σημείο. Τούτου λεχθέντος. Δεν είναι εύκολο να επιτύχει αυτό το εγχέρμα, γιατί όπω είπε και ο κύριο Σταμασούρ και η κυρία Γκουρμάη, υπάρχουν πολλά πολιτικά θέματα και τεχνικά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την αριθμητική επανάσταση που έφερε την Ευρώπη στο να έχει 27 κράτη και τις δυσκολίες οργανωτικές που συνάπτονται με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι είναι μια πρωτοβουλία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι το δικαίωμα αυτό αφορά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα υποφελθούν όλοι από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο από αυτό το οποίο λέει η συνθήκη και αυτό που εμείς διεκδικήσαμε να ενσωματώσουμε στη συνθήκη. Είναι επίσης προφανές, το είπε και ο κύριος Γουόλς, ότι πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν όχι, αν δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δράσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε την εντύπωση και την προσδοκία ότι η πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να γίνουν και από τη συγκριτική μελέτη του δικαίου στα κράτη-μέλη δεν βλέπω κάτι που να με κάνει να πιστεύω ότι με μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να τροποποιηθεί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η ίδια συνθήκη περιλαμβάνει διατάξεις για την ε, τροποποίηση της ίδιας αυτής της συνθήκης. Να συγκληθεί μια συνέλευση λοιπόν για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει νόημα λοιπόν από πολιτική έποψη να θεωρήσουμε ότι μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αλλάξει συνθήκε και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ από την αρχή. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω του δύο εισηγητέ και τον κύριο Χάφνο και και την κυρία Γουάλη για τι προσπάθειε που κάνανε να γίνει φιλική προ του πολίτε αυτή η διαδικασία, να διευκολύνει τη διαδικασία και να είναι ώστε να το λιγότερο επαχθεί αυτή η διαδικασία για του πολίτε προσκρούμε πάντα στο δίλημα του πώς θα συνδυάσουμε και θα παντρέψουμε την ελευθερία με την ασφάλεια. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο, και το λέω γιατί επίκειται και η διαπραγμάτευση των συντονιστών με το Συμβουλίο, υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Όλο αυτό το θέμα της συλλογής και της επικύρωση των υπογραφών πρέπει να γίνει από τα κάτι μέλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εναλλακτική λύση γι' αυτό. Αλλά ειλικρινά Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο εάν τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα κάνουν <clears throat> την επαλήθευση να τους επιβάλλουμε εμείς τους κανόνες βάσει των οποίων θα πρέπει να το πράξουν. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωσης εν τη πολυμορφία. Πρέπει να βασιστούμε στην αγαστή συνεργασία, στην συνεργασία που είναι πιστή στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κράτος μέρος που δεν θα εφαρμόσει τους κανόνες με το πνεύμα αυτό. Μία ομογενοποίηση θα ήταν πάρα πολύ πολύπλοκη. Επίσης, <clears throat> θα πρέπει να δώσουμε μια σοβαρότητα στο εγχείρημα αυτό, να το διευκολύνουμε αφενός, αλλά να το επενδύσουμε και με σοβαρότητα. Θυμάμαι αυτά που έλεγε η κυρία Τέιν που λέ, ομιλούσε για κάποιο Χάν Σμιτ, ο, οποίος να υπογράφει κάποιος ω Χάν Σμιτ από το Βερολίνο. Ποιο είναι ο Χάν Σμιτ, πόσοι Χάν Σμιτ μπορεί να ζουν στο Βερολίνο. Να υπάρχει λοιπόν η φιλική προς τους πολίτες προσέγγιση, αλλά να υπάρχει και μια ελάχιστη σοβαρότητα. Τέλος, σε τεχνικό επίπεδο είναι τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να ρυθμίσουν αυτό το θέμα σε τεχνικό επίπεδο. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη λοιπόν και φυσικά θα πρέπει να διατηρήσουμε και μια σχέση εμπιστοσύνη με τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με τον κύριο Ντάφ για κάτι που είπε. Το θέμα των υποχρεωτικών δημοσίων ακροάσεων θα δημιουργήσει ένα τεράστιο βάρο. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να είναι απαραίτητο, μπορεί να μην είναι. Μπορεί η Κομισιόν να θεωρήσει ότι είναι καλή πρωτοβουλία και να κάνει αυτή την ακρόαση ούτω ή άλλω. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια πρωτοβουλία που να είναι φιλική προς τους πολίτες, πρέπει να είναι φιλική και προς την Κομισιόν, να μην οδηγήσει σε υπερβολικές υποχρεώσεις για την Κομισιόν. για την ε, θέση σε εφαρμογής. Κατανοώ το επιχείρημα του κ. Κασίνη. Η ευαισθησία μου μου λέει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει κάτι τέτοιο και τα κράτη-μέλη καθυστέρησουν πάρα πολύ, αυτό δεν θα είναι πρόσφορο. Πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Και το είπε ήδη ο κύριος Κασίνη. Η Κομισιόν μας δίνει 6 με 9 μήνες για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πληροφορική για τι υπογραφέ και τα κάτι μελιθαίνουν 12 μήνε, κάπου πρέπει να, βρεθούμε, να βρεθεί μια λύση στη μέση. Για την Κοντέσα Τούν και Χόχενστάιν, που έθεσε ένα ερώτημα. Και λέει για το αν η, έθεσε το ερώτημα του αν οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Ακούσαμε τις ε, απόψεις υπέρ και κατά για το θέμα αυτό πιστεύω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Όχι ότι δεν είμαστε πολίτες, είμαστε, αλλά έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να παρουσιάσουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες. Και πιστεύω πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. <clears throat> Είναι γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Αυτό Κοινοβούλιο υπάρχουν συνάδελφοι που ξεκινήσανε να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες ή τουλάχιστον να τις ε, υποστηρίζουν δημιουργείται μια σύγχυση ρόλων που εγώ θα προτιμούσα να την, ε, να την αποφύγουμε. Αυτό μπορεί να, μου φαίνεται, να μπορεί να σας φαίνεται κάπως αφελές, αλλά εγώ θα ήθελα η πρωτοβουλία πολιτών να μην ξεκινάει από αυτούς που είναι οργανωμένοι πολίτες, αλλά από τους απλούς πολίτες. Για το ΕΛΚ λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε σκεφτεί πολύ τις τροπολογίες αυτές οι οποίες ε, κατατέθηκαν και νομίζω ότι καταδεικνύουν και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουμε για το θέμα αυτό. <clears throat> Πιστεύω ότι με την ε, αυριανή ψηφοφορία θα δώσουμε στους εισηγητές μια εντολή για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν. Θα τους δείξουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη μας. Είναι σημαντικό όμως να έχουν και μια <clears throat> ευελιξία σε σχέση με την πολιτική δράση τους. Ο κ. Λαμασού γνωρίζει πολύ καλά το σύστημα του μπαλοτάζ των δύο γύρων στη Γαλλία και σε άλλε χώρε. Λέει ότι στον πρώτο γύρο λέει κάνει ό,τι θέλει, ψηφίζει ό,τι θέλει. Στο δεύτερο γύρο παίρνει την πραγματική απόφαση. Το αφήνω πάντω στην ε, κρίση των εισηγητών για το πώς θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην εντολή που θα του δώσει η Επιτροπή μα αύριο. Εγώ τονίζω και πάλι ότι πρέπει αύριο που θα ψηφίσουμε να τονίσουμε ότι είναι μια σημαντική μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Κύριος Γκρότε, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, είναι τα γενοφάσκια της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών που γιορτάζουμε. Αυτό είναι ένα γιγάντιο βήμα και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν φανταζόμασταν εμεί στο παρελθόν ότι θα μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε σε μια στιγμή που θα υπάρχει η άμεση συμμετοχή των πολιτών στο πολιτικό γύρνισθε. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και του δύο εισηγητέ γιατί έχουν κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και ίσως έχω εκνευρίσει μερικές φορές την κυρία Γκουρμάη με τις προτάσεις που έχω υποβάλει. Παρ' όλα αυτά έδειξε μια μεγάλη εγκαρτέζη και υπομονή μαζί μου και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και την ευχαριστώ λοιπόν. Ο στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι να καρποφορήσει αυτή η πρωτοβουλία και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο γεγονός αυτό ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι εκτεταμένη πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συλλέγονται και οι πληροφορίες και οι υπογραφές μάλλον ε, επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Και έχουμε αναφέρει ότι όταν κανείς υπογράφει κάτι δεν πρέπει να αναφέρει το αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλοι είναι έτοιμοι να υπογράψουν, αλλά άμα αρχίσουμε να ρωτάμε τους πολίτες για δώστε μας τα στοιχεία σας, της αστυνομικής σας ταυτότητα, αυτό αποτρέπει πάρα πολλούς. Η υπόθεση με το Χάν Σμιτ, το παράδειγμα αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, Ε, που μπορεί να ζουν δύο Hans Schmidt στο ίδιο σπίτι στο Βερολίνο, αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Σε σχέση με τη διαδικασία, η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας αν υπάρχει η δυνατότητα ανθρώπων έξω από τους θεσμικούς φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απόψεις για το πώς θα πρέπει να ζει η Ευρώπη, τι ε, θα πρέπει να κάνει. Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε κάτι το οποίο είναι έξω από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος όμως θα πρέπει να είναι ακόμα και οι μη πραγματοποιήσιμες προτάσεις να μπορούν να τύχουν κάποιες ακρόασεις. Δηλαδή να έχουμε κάποια σκέψη για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ιδέες. Η κοινωνία των πολιτών και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς πάντα έχουμε κάνει προσπάθεια να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όταν υπάρχουν ευρείες συζητήσεις και να μην είναι μονάχα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρόντες που έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην νομοθετική ε, διαδικασία. Εάν εμείς θέλουμε να κάνουμε πολιτική, εδώ είναι ο χώρος που πρέπει να το κάνουμε. Όταν όμως τώρα μιλάμε για κόμματα που μπορεί να μην έχουν μια εκπροσώπηση παραγωγής χάρη μέσα σε μια βουλή, τα κόμματα, τα συνδικάτα και οι μη, μη κυβερνητικές οργανώσεις ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια. Εγώ υποστηρίζω να υπάρξει διαφάνεια για τη δρόση όλων αυτών. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε κόμματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Στα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι <clears throat> ανήκουν στην ε, κοινωνία των πολιτών και δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την ε, δυνατότητα πρωτοβουλίας ε, πολιτών. Υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο τρόπο, τρόπο να το παρακάμψει αυτό κανείς μέσα από συνδικάτα ή άλλους φορείς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι Πρέπει να διατηρήσουμε την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, την υποστήριξη και την χρηματοδότηση. Και να μην πούμε επομένως ότι αποκλείονται τα κόμματα, τα κόμματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Για μας είμαι σύμφωνος, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εδώ πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, δεν υπάρχει το αντίστοιχο του σε παγκόσμια κλίμακα Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ απόψει τώρα για τα πιο λεπτομεριακά σημεία, αλλά αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα είναι κάτι το συναρπαστικό αν τελικά καρποφορήσει αυτή τη διαδικασία και έχουμε αυτό το εργαλείο της ε, πρωτοβουλίας πολιτών. Ευχαριστώ και πάλι στους ηγητέ. Ευχαριστώ. Ich möchte auch gerne noch mal einige Punkte και εγώ θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν για το χρονοδιάγραμμα. Ε, είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Υποστηρίζω λοιπόν τον εισηγητή, τον πρόεδρο μάλλον, για το γεγονό ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένα χρόνο για τα κάτι μελη για να εφαρμόσουν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένου ότι μέσα σε έξι μήνες μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία απαιτείται στα κράτη-μέλη. Και επίσης μπορεί να υπάρχουν και ορισμένε προδιαγραφές σε επίπεδο ποινικού δικαίου οι οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορεί να εμποδίσουν τους ε, συντάκτες, τους προτείνοντες μια πρωτοβουλία να λειτουργήσουν. Ε, στην περίπτωση της ε, Γερμανίας, εάν είναι άκαρτη μια πρωτοβουλία πολιτών, πάντα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη πρωτοβουλία. Αλλά υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος να δημοσιοποιηθούν υπογραφές και να πουληθούν ακόμα σε ιδιωτικούς φορείς. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν λοιπόν οι απαραίτητοι κανόνες οι οποίοι θα θεσπιστούν και έξι μήνες μπορεί να μην είναι επαρκείς για να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες διασφαλίσεις. Θέλω επίση να υποστηρίξω αυτά που λέει η κυρία Τούν ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν οι κοινοβουλευτικοί στην Οργανωτική Επιτροπή, είτε είναι ευρωβουλευτέ είτε εθνικοί βουλευτέ. Είμαι τελείω εναντίον μια τέτοια ρύθμιση που θα επέτρεπε κόμματα ή συνδικάτα ή νομικά πρόσωπα να είναι τμήμα της Οργανωτικής Επιτροπής. Η πρωτοβουλία πολιτών οι πρόσωπα. Εγώ δεν θέλω να βρεθώ στην κατάσταση να ελέγξω αν ένα νομικό πρόσωπο έχει, έχει εκπροσωπηθεί νομο, ας σε μια οργανωτική επιτροπή. Το πρόβλημα με τα νομικά ε, πρόσωπα είναι ότι το Προεδρείο, οι εκπρόσωποι <clears throat> πολλές φορές αλλάζουν και αλλάζουν συνέχεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς ότι τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανόνες για την εκπροσώπηση από ένα πρόεδρο, από ένα διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως θα είναι επαχθής η διαδικασία για κόμματα ή για συνδικάτα όταν πρέπει κανείς να κάνει μια τέτοια εκστρατεία. Δεν πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή παρά το γεγονό ότι μπορούν να υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία. Ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον οι πολίτε τρίτων χωρών που είναι μόνιμα κάτοικοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την Οργανωτική Επιτροπή. Η φιλελεύθερη ομάδα δεν έχει μια ενιαία άποψη για το θέμα αυτό, αλλά εμείς ως ε, γερμανική συνιστόσα της Άλντε θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπορούν να υπογράφουν μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζεται με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολίτης μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει πραγματικό πρόβλημα για το κατά πόσο ένα άτομο ε, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει γιατί πρέπει να γίνει ο έλεγχος του αν πράγματι μένει μόνιμα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Επίσης, ξαφνικά αν έρθει ένα εκατομμύριο Κινέζων στην, ε, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να κάνουν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που έχει να κάνει με την Ευρώπη. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει λογική να μπορούν οι πολίτες της, οι μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζουν, να υπογράφουν μια πρωτοβουλία. Για την οριακή ηλικία εγώ υποστηρίζω όπως ο πρόεδρος της την ηλικία των 18 ετών που συνάδει με την ε, παράδοση στα κράτη-μέλη και φυσικά πιστεύω ότι αν δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση θα πρέπει να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως θα ήταν χρήσιμο να υποστηρίξουμε μια ηλικία μέσα από αυτή την πρωτοβουλία 16 ετών για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής Αναφορών και αυτό το οποίο είπε πει και ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, ότι δεν πρέπει να οργανωθεί μια ακρόαση για τις πρωτοβουλίες από την Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, αλλά μια λύση θα ήταν να το πράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη Επιτροπή Αναφορών. Τώρα, αν πρέπει να είναι αυτή η Επιτροπή ή όχι, αυτόν είναι δευτερεύον. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να οργανωθεί μια ακρόαση από αυτούς που πιστεύουν ότι η Κομισιόν δεν έχει πράξει όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει και οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πιο κοντά στους πολίτες και να δώσουν τη δυνατότητα να ακουστεί αυτή η πρωτοβουλία στα και στα μέσα ενημέρωση και επομένω να υπάρξει μια πιο επίσημη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Ευχαριστώ. Τρία σχόλια πολύ σύντομα. Πολλοί μίλησαν για το ποιο μπορεί να υπογράψει την πρωτοβουλία των πολιτών. Αν διαβάσουμε τη συνθήκη, λέει θα πρέπει να είναι υπήκοοι ενό μεγάλου ρυθμού κρατών μελών. Το να το διευρύνουμε περαιτέρω νομίζω ότι αντιβαίνει σε αυτό που συμφωνήσαμε στα πλαίσια τη συνθήκη. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα πιο θετικό επιχείρημα. Μονίμω ε, πρέπει να σα πω μάλλον ότι στη συνθήκη του Μάστρεχτ ε, δημιουργήσαμε την έννοια τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ήταν μια μεγάλη ιδέα που. Και μάλιστα μέσω αυτή τη πρωτοβουλία θα δώσουμε ε, σάρκα και οστά στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια θα την κάνουμε πιο ελκυστική στον Ευρωπαίο πολίτη. Πόσοι γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ε, ξέρουν τι σημαίνει η συμμετοχή τους στις εκλογές κτλ. Αλλά για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια τι γνωρίζουν. Νομίζουμε ότι μπορούμε να διαφημίσουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια μέσω της ε, πρωτοβουλία των πολιτών. κάτι που θα ήθελαν και οι συντάκτες τη ε, συνθήκη του Μάστρικ αντί να το λέμε αρνητικά, να λέμε να περιορίσουμε το α και το β, ας το πούμε θετικά. Ε, ας δώσουμε αυτή την ε, εξήγηση. Γιατί περιοριζόμαστε στους υπηκόους των κρατών μελών. Ε, και μια και το λέμε, ε, το ονομάζουμε, ονομάζουμε αυτή την πρωτοβουλία, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων ε, υπηκόων, των Ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτούς. Έπειτα, από πόσα κράτη-μέλη θα πρέπει να προέρχονται οι υπογράφοντες. Θα πρέπει να είμαστε απλώ συνεπεί. Όταν μιλάμε για ενισχυμένη συνεργασία, στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνουμε πολλά κράτη-μέλη. Ε, αυτό ε, εν συνεχεία μεταφράστηκε σε συγκεκριμένο αριθμό μελών στη συνθήκη. Δεν θα έχει νόημα σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα, ε, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην ενισχυμένη συνεργασία, να έχουμε μικρό αριθμό κρατών μελών θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. Και έπειτα, με αυτό το πρόβλημα, τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα που έχουμε, αν οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωβουλευτέ, οι εθνικοί βουλευτέ έχουν το δικαίωμα να προσυπογράψουν την πρωτοβουλία των πολιτών. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα και των μεν και των δε, αυτών που λένε ότι εμεί δεν πρέπει γιατί έχουμε άλλα μέσα, α πούμε άλλα μέσα για να συμμετάσχουμε στην πολιτική διαδικασία, στο πολιτικό γίγνεσθε. Αλλά καταλαβαίνω και αυτός που λένε ότι μα και εμεί το κάτω-κάτω πολίτε δεν είμαστε. Νομίζω ότι η... ο συμβασμό που ακούστηκε από τον Αλά είναι καλό. Θα υπάρξουν πολλέ περιπτώσει όπου κάποιοι από εμά, κάποιοι από του εθνικού βουλευτέ θα εμπλακούν στη διαδικασία. Ακόμα και τώρα. Και ίσω και εσεί έχετε αντίστοιχη εμπειρία. Ε, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος μας πλησιάζει και μας λέει πώς να το κάνουμε, ας πούμε, μπορείτε να μας βοηθήσετε, ε, ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν στις επιτροπές σας κτλ. Και ούτως ή άλλως ο ρόλος μας είναι να τους ε, συμβουλεύσουμε. Για λόγους διαφάνειας λοιπόν, όσοι εμπλέκονται και βοηθάνε τους πολίτες να οργανωθούν, αν μπουν στην Οργανωτική Επιτροπή και μόνο, και μόνο για λόγους διαφάνειας δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Γιατί έτσι στέλνουμε και ένα μήνυμα στους πολίτες ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι και άλλες οδοί για να κάνει κανείς πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε και διαφάνεια, εμπλέκονται όλοι, γιατί οι εθνικοί βουλευτές, σας το λέω από τώρα, θα εμπλακούν ούτως ή άλλως. Και απ' την άλλη ο κόσμος θα ξέρει ότι οι ψήφοι, του, οι ψήφοι των βουλευτών ε, δεν μετράνε. Απλώς εμφανίζονται τα ονόματά τους στην Οργανωτική Επιτροπή. Μερικές φορές βοηθάει τον εμφανίζονται αυτά ονόματα. Ε, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, προσανατολίζεται με βάση αυτά τα ονόματα. Ευχαριστώ κύριε Ταρκόσκη. Κυρία Γιατεμάκη. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. try to be brief. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. δασά σημεία θα υπογραμμίσω. Ευχαριστώ καταρχάς τους εισηγητές. Κάνανε μια μεγάλη, μια πολύ σημαντική προσπάθεια, την κάνανε αυτοί και εμείς. Και εμείς τώρα στο τέλος θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντική όλη η προσπάθεια για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να τα καταφέρουμε. Το να αποτύχουμε τώρα θα ήταν πολύ άσχημο για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ άσχημο για τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτή την ιστορία. Άσχημο και για το Κοινοβούλιο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά και για την Επιτροπή μας. Τώρα, συμφωνώ ότι θα πρέπει η προσπάθεια, θα πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να είναι φιλική προς τους πολίτες. Το λέμε όλοι αυτό. Τι σημαίνει όμως αυτό. Για μένα, Φερρυπίν, τι σημαίνει. Ότι θα πρέπει να, είναι η... θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσφύγουμε στο ΔΕΚ και στο διαμεσολαβητή σε περίπτωση που υπάρχει κακή διαχείριση. Σε περίπτωση κακοδιαχείρισης Μπορεί να υπά... Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ελπίζω να μην υπάρξουν τέτοιε περιπτώσει. Αλλά αυτοί που δούλεψαν για την πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω βέβαια ότι μπορούν να πάνε στο δικαστήριο, αλλά καλό θα ήταν να το γράψουμε κιόλα. να το πούμε ξεκάθαρα στην έκθεση, ούτω ώστε να το βλέπουν οι πολίτε, να το βλέπουν όλοι. Εμεί το ξέρουμε, αλλά δεν το ο κάθε πολίτη. Δεύτερον, αντίθετα από τη Γερμανίδα στην αδελφό μου, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι όσοι διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν δυνατότητα να υπογράψουν μια πρωτοβουλία. Είναι θέμα ελευθερίας λόγου, ελευθερίας του συνέρχεστε. Είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει σε όλους. Σε όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το δικαίωμα είναι διαφορετικό από το δικαίωμα στις εκλογές, το δικαίωμα του να ψηφίζει κανείς. Έχω και πρακτικά επιχειρήματα να σας αναφέρω. Φανταστείτε ότι υπάρχουν δύο, τρία, πέντε άτομα που σκέφτονται να προσυπογράψουμε την πρωτοβουλία. Ας την υπογράψουμε, λέμε. Κάποιοι από αυτού μπορεί να είναι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι όλη παρέα. Δεν είναι όλη παρέα υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιε διακρίσει μεταξύ πολιτών και μη πολιτών. Τρίτο σημείο, που μπορεί να φαίνεται ίσονο σημασία, έχει να κάνει με την ε, διάκριση, με διακριτική μεταχείριση. Πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν. Είναι πολύ σημαντική η διασφάλιση αυτού του δικαιώματος. Γι' αυτό πρότεινα λοιπόν να αναφέρουμε εδώ και τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες. Γιατί και οι δικές τους φωνές πρέπει να ακουστούν. Εφόσον λέμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τους πολίτες με ισονομία, τους πάντες με ισονομία, θα πρέπει να το γράψουμε αυτό και εδώ. Για τις ακροάσεις, συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι μπορεί να αποβεί σημαντικό, μπορεί και όχι. Εδώ διοργανώνουμε πολλέ ακρόασει. Αρκεί να προτείνει ένα, δύο, τρει. τη διεξαγωγή μιας ακρόαση. Αν έχουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει να διοργανώσουμε μια ακρόαση. Ακόμη και αν δεν προκύψει νομοθέτημα, ακόμη και αν δεν προκύψει οδηγία ή κανονισμός από αυτές τις υπογραφές τουλάχιστον να κάνουμε μία ακρόαση για να ακούσουμε αυτές τις γνώμες. Δεν ξέρω βέβαια αν οι επίτροποι ή κάποιοι άλλοι μεγαλόσχημοι έχουν άποψη για, το, για αυτό το θέμα. Το θέμα μάλλον μου φαίνεται πιο πολιτικό από οτιδήποτε άλλο, από νομικό ή τεχνικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Έχω, έχω τι εξή παρατηρήσει πρώτα-πρώτα όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων σε αυτή τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη ότι πάρα πολλά κόμματα στην Ευρώπη δεν εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Και ίσω δεν είναι και τόσο έξυπνο του να του αφήσουμε απ' έξω όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Σε σχέση με τι δυνατότητε που έχουμε εμεί ω βουλευτέ. Γιατί ξέρετε, στην Ιταλία έχουμε ένα σωρό κόμματα που, που, που, που είναι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω δεν έχει νόημα να του αφήσουμε έξω από αυτή τη διαδικασία τη πρωτοβουλία των πολιτών. Κατά δεύτερο λόγο, έχω κάπως προβληματιστεί, όχι τόσο για το τι γίνεται, οπότε είναι παραδεκτή μια πρωτοβουλία, αλλά όταν είναι απαράδεκτη, τι γίνεται τότε. Και κοιτάξτε τις ε, ευρωπαϊκές συμβάσεις ε, και τα σχετικά. Υπάρχει συνήθως κάποιο ένδικο μέσο. Είναι βασικό δικαίωμα και λέει εδώ περί Ευρωπαϊκή Τροπή ότι δύναται να κηρύξει το απαράδεκτο. Τότε τι κάνει κανείς. Σε δεύτερο βαθμό, πού πάει κανείς δεύτερη ανάγνωση, πέστε το όπως θέλετε, πέστε το εγώ έχω μια τροπολογία. Δηλαδή, να μην περάσει το 144 ότι όταν επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει μια πρωτοβουλία, μια πρόταση, τότε εμείς να το ξανασυζητούμε. Αν θέλουμε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σκεφτώ μια που εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους. Άρα αυτό θέλω να το πω, να το λάβει όψη ο κύριος Λαμασούρ. Τι λέτε κύριε Λαμασούρ επ' αυτού. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα ας πούμε έφεσης προσφυγής εάν ε, η Επιτροπή απορρίψει μια πρωτοβουλία και εν τη περιπτώσει πού αλλού να ζητηθεί σε δεύτερο βαθμό η περίπτωση παρά εδώ, εδώ και ένα χρόνο. το κουβεντιάζουμε. Εδώ είναι ο σωστός τόπος. Και σε σχέση και με την εντολή που έχουμε λάβει εδώ είναι το πιο σωστό φόρουμ σε δεύτερο βαθμό να συζητηθεί το παραδεκτόν. Επομένω, πρώτον, συμμετοχή πολιτικών κομμάτων και δεύτερον, κατά πόσον οι συνεισηγητές θα πρέπει να δώσουν αυτό το δημιουργείο για να το αναγνωρίσουν τους του υπογράψοντες μία πρωτοβουλία. Αυτά. Χωρίς μικρόφωνο Πρόεδρος. Δίνει το λόγο στον επόμενο. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Και εγώ να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η δημόσια συζήτηση. Υπάρχει μια διάσταση η οποία κάνει αυτή τη δημόσια συζήτηση πάρα πολύ επιθυμητή είναι το θέμα της προβολής στα μέσα ενημέρωσης και της διάδοσης της, ε, μετα, της, ε, του να γίνει γνωστό αυτό το θέμα. Είναι ένα είδος κατάστασης που αρέσει ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωση να παρουσιάζουν τέτοιες προτάσεις και αυτό είναι μια ευκαιρία να γίνει ευρύτερα γνωστή μια πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το τεκμήριο του ενδιαφέροντος ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια ακρόση και αυτό να είναι στην κρίση των ε, οργανωτών μιας πρωτοβουλίας. Για την επαλήθευση τώρα των, των υπογραφών θα πρέπει να είμαστε προς την κατεύθυνση της αυστηρότητας. Υπάρχει κίνδυνος αν είναι υπερβολικά εύκολο να παρα, ε, χαράξει κανείς τις υπογραφές ας πούμε άλλων. Αυτό θα θέσει υπό αμφιβόλο και θα ουσιαστικά θα μείωσει το κύρος αυτής της πρωτοβουλίας. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν στοιχεία σε ταυτότητες θα πρέπει να δείχνει κανείς αυτό το, αυτό το έγγραφο το επίσημο και στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχει κανείς ταυτότητα μπορεί να δείχνει ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ή νερό. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι το να έχουμε μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που υποστηρίζω, αυξάνει την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλουμε να εξάρουμε, το ρόλο του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλαμε να το ονομάσουμε διαφορετικά, το ονομάζαμε διαφορετικά. Πρέπει να είναι κάτι που συνάπτεται με την έννοια της ηθαγένεια της ευρωπαϊκής Για τον κύριο Νταφ, ο οποίος αναφέρθηκε για τους ε, Ρώσους στη Λετωνία. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, οι Ρωσόφωνοι αν θέλετε περισσότερο, στην ε, Εστονία και στην Λετωνία έχουν υπηκότητα και υπάρχουν περίπου 300.000 Ρώσοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως ο κ. Ντάφ θεωρεί ότι και αυτοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία πολιτών. Πριν, το δώσω, πριν λόγο στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, θα ήθελα να παρέμβω κι εγώ εκ νέου. Λάβετε υπόψη σα ε, ότι αύριο δεν θα είμαι παρόν. Οπότε δικαιούμαι. Ένα γύρο ακόμα. Ε, η συζήτηση ήταν, πολύ πλούσια. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν ε, τι εξή παρατηρήσει. Το άρθρο 1.14 λέει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι ένα εκατομμύριο. Τώρα, το να δεχτούμε μη πολίτε ε, να υπογράφουν και αυτή την ε, πρωτοβουλία θα ήταν παραβίαση τη συνθήκη. Ένα εκατομμύριο πολίτε, λέει η συνθήκη. Δεύτερον, το θέμα του, των έξι μηνών ή του ενός χρόνου. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά προβλέπεται η Επιτροπή μέσα σε έξι με εννέα μήνες να εκπονήσει τους κανόνες για την καταχώρηση και την ψηφοφορία. Ε, μέσω βίντεο διάσκεψης. Ε, είναι κάτι πολύ καινοφανές αυτό. Εγώ δεν πιστεύω πολύ σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι πουθενά σε καμία χώρα δεν προβλέπεται τέτοια τηλεματική ψηφοφορία. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα η Κομισιόν να εκπονήσει αυτό το σύστημα για να αποφασίσει μετά πώς θα εφαρμοστεί στις επιμέρους ε, χώρες. Ε, η Κομισιόν έχει εννιά ε, μήνες. Πώς μπορούν να τα καταφέρουν τα, κράτη-μέλη μέσα σε έξι μήνε να οργανωθούν να οργανωθούν και να εφαρμόσουν ένα τόσο καινοφανέ και περίπλοκο σύστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ε, όχι 6 μήνε, αλλά ένα χρόνο για τα κράτη-μέλη. Τρίτον, το είπαν κι άλλοι, το τονίσω κι εγώ. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα της, ε, της, ε, του ιδιονόματος, αλλά της αλλά και της ε, παραποίησης των ε, υπογραφών. Επίσης, μπορεί κάποιος να πάει να βάλει το όνομα κάποιου που δεν έχει ιδέα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα με την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να επαληθεύεται το αυθεντικό της ε, υπογραφής. Μπορούμε να το κάνουμε και δειγματοληπτικά. Να επαληθεύσουμε ότι το γνήσιο της υπογραφής για ένα μεγάλο αριθμό υπογραφόντων. Να έχουμε ένα μεγάλο δείγμα. Ε, εάν οι πολίτες δεν θέλουν κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι δεν πιστεύουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Για το τελευταίο θέμα. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι αυτή. Τη δυνατότητα προσφυγής. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που θέλουν να δώσουν την πρωτοβουλία αυτή, να συναρτήσουμε την πρωτοβουλία αυτή με τη δυνατότητα προσφυγής. Δυνατότητα προσφυγής στο 10. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα τα δουν όλα αυτά οι συγγητές. Αλλά η δική μας επιτροπή, η οποία ασχολείται με τις συνταγματικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει πολύ σύντομα να επιλύει προβλήματα Ξέρετε ότι πολύ γρήγορα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Φανταστείτε, ε, εμείς δουλεύουμε πολύ, δουλεύουμε αμελητή, αλλά φανταστείτε πώς δουλεύει το ΔΕΚ, που, έχει, που κατακλείσεται, κατακλείσεται από υποθέσεις. Υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με την προσφυγή πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό το θέμα ε, και σκεφτείτε και τις σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Η Κομισιόν ιδιαίτερα αισιόδοξη, ε, ιδίω μετά από την συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων που έχει λάβει η χώρα και πιστεύει ότι μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται επιτάπητος. Τέσσερα σημεία τα οποία είναι κάπως προβληματικά για μας θα ήθελα να αναφέρω και θέλω να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για το θέμα της προσφυγής, δυνατότητας προσφυγής. Το πρώτο θέμα που θέλω να συζητήσω είναι το θέμα της ενδεχόμενης δημόσιας ακρόασης. Η Κομισιόν συμφωνεί περισσότερο με αυτούς όπως ο κύριος Ντάφ και ο κύριος Μέντες Δεβίγο οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση για την οργάνωση αυτής της ε, ακρόασης εάν το Κοινοβούλιο επιμένει να υπάρχει η εγγύηση μια νομικής επιταγής για αυτή την ε, ακρόαση. Η Κομισιόν έχει τονίσει ότι δεν πρέπει να είναι η Κομισιόν η οποία θα οργανώσει κάτι τέτοιο, αλλά το Κοινοβούλιο, γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να, να έχει το κίνδυνο να κατηγορηθεί για κακοδιοργάνωση μιας ακρόασης, ότι δεν έχει οργανώσει σωστά την, ε, την ε, ακρόαση για να πετύχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ευνοϊκό, εφόσον η Κομισιόν υποτίθεται ότι είναι η αρμόδια για την έγκριση. Για τις γλώσσες επίσης πρέπει να κρατήσουμε την ε, σαφήνεια της αρχικής πρότασης που λέει ότι το αρχικό, η αρχική καταγραφή πρέπει να γίνει μονάχα σε μία γλώσσα και επί τη βάση αυτής η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει τον έλεγχο και μόνο όταν υπάρξει η επικύρωση καταγραφής τότε φυσικά θα πρέπει να είναι δυνατόν να δοθούν στην Κομισιόν και οι μεταφράσει σε άλλες γλώσσες και η Κομισιόν θα τις θέσει στο κατάστοιχο ώστε να μην γίνεται εξ αρχής περίπλοκη η όλη ιστορία της καταγραφής. Θέλουμε να κρατήσουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα. Το ίδιο αφορά το νέο άρθρο 20β για την αρρωγή η οποία παρέχεται. είπαμε ότι θα προβλέπετε κάποιο help desk, μια βοήθεια, μια υποστήριξη για να μπορούν να καταγράφονται οι πρωτοβουλίες και για να διευκρίνονται διάφορα σημεία με τους οργανωτές μιας πρωτοβουλίας. Μας φαίνεται όμως πολύπλοκο και επικίνδυνο να υπάρξει και η δυνατότητα μιας νομικής ε, συζήτησης η οποία θα είναι υποχρεωτική. Νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να καθορίσει τι θα κάνει, να το διευκρινίσει με μία ανακοίνωση και αν το Κοινοβούλιο θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει περαιτέρω ε, ρήτρα, θα, μπορεί, θα μπορούσε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορούμε να πούμε απλώς μια ρήτρα ότι θα υπάρξει υποστήριξη από την Κομισιόν στο κείμενο και εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει σε ένα αυτόνομο άρθρο, αλλά στο ίδιο το άρθρο 4, αυτό που ανέφερε ο κύριος ε, Λαμασούρ, για τη διαδικασία καταγραφής, εκείνη ίσως τη στιγμή που θα πούμε ότι θα υπάρχει μια δυνατότητα υποστήριξης από την πλευρά της Κομισιόν. Τέταρτο σημείο, η ρήτρα αναθεώρησης. Θα κάνω εδώ μια έκκληση να προσπαθήσουμε να είμαστε νυφάλοι και να διατηρήσουμε την απλότητα. Κάθε τρία χρόνια μπορεί να... Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο χρονικός ορίζοντας. Εμείς είχαμε πει κάθε πέντε χρόνια, αλλά αναθεώρηση κάθε τρία χρόνια αυτό είναι υπερβολικό. Έτσι και αλλιώ τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για όλους στις ιστοσελίδε, Τα αποτελέσματα όλων των πρωτοβουλειών, το πόσε ε, ευδοκίμησαν και ποιε όχι, σε πόσα απήντησε η Κομισιόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει η νομική υποχρέωση επανεξέτασης κάθε τρία χρόνια. Και είδαμε και στο Συμβούλιο επίσης. Ορισμένοι να θέλουν να γίνεται μία επανεξέταση στο α και β σημείο για το επιγραμμικό σύστημα, για τις επιτροπές πολιτών, για τα θέματα διαφάνειας κτλ. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα τεράστιο κατάλογο ο οποίος θα υποβαθμίσει λιγάκι το έργο μας γιατί αν έχουμε πάρα, πολύ, ε, πολλά σημεία που πτήθανε στον κατάλογο αυτό γεννά και αμφιβολίες στο πνεύμα των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε ένα απλό τρόπο ε, επανεξέτασης, να δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα. Μια τελευταία διευκρίνηση για το θέμα του, της δυνατότητα προσφυγής που αναφέρθηκε. Βέβαια, ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέσα στο κείμενο. Εάν ο πολίτης θεωρεί ότι υπήρξε κακοδίκηση από την πλευρά της Κομισιόν, υπάρχει πάντα δυνατότητα να απευθυνθεί στο διαμεσολαβητή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και οι εθνικοί μεσο... διαμεσολαβητές μπορούν να παρέμβουν αν οι εθνικέ αρχέ δεν κάνουν σωστά την επαλήθευση των υπογραφών παραδείγματο χάρη. Αυτές είναι ρυθμίσει οι οποίε ήδη ισχύουν. Και εάν δεν υπάρξει καταγραφή μια πρωτοβουλία σε ένα μητρό, εκεί προφανώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απλώ έχουμε την τροπολογία που λέει ότι η Κομισιόν όταν απορρίπτει μια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να πληροφορεί του πολίτε για τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή του. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση, αλλά δεν πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά στοιχεία λεπτομεριακά στο κείμενο για την προσφυγή, την δυνατότητα προσφύγή. Αυτά δεν χρειάζεται να είναι στο κείμενο το ίδιο. Ευχαριστώ. Eh, ah, eh, Έχουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να μιλήσει. Βεβαίω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα σας αναφέρω ένα δύο θέματα. πρώτα πρώτα θα σα πω ότι για μένα τα μεγάλη τιμή να παραστώ σε αυτή τη συζήτηση και να ακούσω την επικοδομητική ανταλλαγή απόψη. Είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο στην κορεπέρ. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω αυτή η επαλήθευση πόσο σημαντική είναι για τα κρατημέλη. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε όσα άκουσα από τις παρεμβάσεις για το πόσο σημαντικό είναι το να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα των κρατών μελών για να αναλάβουν το καθήκον της επαλήθευσης μια που έχουμε τόσα πολλά διαφορετικά συστήματα. Δεν μπορεί να γίνει εναρμόνιση βροχυπρόθεσμα, έτσι απλά. Και μετά από μακρές συζητήσεις στην ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο δουλέψαμε πολύ με στόχο την απλούστευση αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι που να τους βολεύει όλους. Επίσης, το θέμα του ορίου ηλικία, διάφοροι από τους αγορητές και αυτοί συμφώνησαν με την κυρίαρχη άποψη στο Συμβούλιο. Ότι το προτιμητέο είναι να υιοθετήσουμε κι εμείς το όριο της ενηλικίωσης. και αυτό να ενταχθεί στο σώμα νομοθετήματος. Κατά τρίτον θα πρέπει να σας επισημάνω το πόσος χρόνος χρειάζεται για την εφαρμογή του κανονισμού. Και σας παραπέμπω στα όσα ακούστηκαν, δηλαδή θα χρειαστεί επιπλέον νομοθεσία και καμιά φορά και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν μπορεί παρά να πάρει πολύ χρόνο. Θα πρέπει στα τα κρατημένα να κάνουν ό,τι πρέπει να το ώστε όλα αυτά να τα επιστατεύσουν. Και γι' αυτό λέμε για αυτό το δεκάμενο. Και τελευταίο, να σας πω για το όπως ακούσαμε έχουμε μια σειρά χωρών που σε αυτή τη φάση πρέπει να συμμετάσχουν στην αναβαθμισμένη συνεργασία, στην συνεργασία τέλο πάντων και χρειάζεται ένα ελάχιστο αριθμό προ τούτο. Εν τρίτον, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα η πρωτοβουλία. Αυτά ήθελα να σα πω και περιμένουμε πώς και πώς να βρεθούμε από αύριο κιόλας στα πλαίσια του τρίμερους διαλόγου. ούτως ώστε όσο γίνεται περισσότεροι να στρατευτούμε για τον κοινό σκοπό και να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Στο μεταξύ έφτασε και ο Επίτροπος, που είναι και Αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής, ο κ. Σεύκοβιτς, τον χαιρετώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που περιπλέξαμε τη συζήτηση για την πρωτοβουλία των πολιτών. δυστυχώς τα θέματα του, τα θεσμικά θέματα του προϋπολογισμού θα πρέπει να τα συζητήσουμε αύριο το πρωί. Ε, θα απαντήσουν κύριε Σεύκοβιτς, άμα σε επιτρέπετε τώρα, οι συγητές και μετά θα σας δώσω τον λόγο. Θα ήθελα λοιπόν η κυρία Γκουρμάη και μετά ο κύριος Λαμασούρ να απαντήσουν και μετά θα σας δώσω τον λόγο κύριε Σεύκοβιτς. Αν μας επιτρέπετε. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε που εσείς και όλο το επιτελείο σας προθυμοποιηθήκατε να συμμετάσχετε και ευχαριστώ τους συναδέλφους τώρα για τα όσα είπαν για τη συμβολή τους και όλοι θέξατε τα ίδια 2-3-4 σημεία τα ίδια σημεία από το κείμενό μας και όπως είπατε αύριο στην ψηφοφορία θα ξεκαθαριστεί αν έχουμε ή όχι πετύχει τη συνένεση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ελπίζουμε κρυστάλλινη να είναι η εντολή που θα λάβουμε σας αύριο. Ευχαριστούμε και τους αδέρφους Κομισιόν και από το Συμβούλιο, οι οποίοι έδειξαν ότι είναι αμύωτο το ενδιαφέρον τους και βεβαίω βοήθησαν ούτω ώστε να καταλήξουμε στις πιο άστοχες συμβαστικέ λύσεις. Ελπίζω να μην έχουμε ευκαιρία να κλείσουμε σε πρώτη το θέμα και όλοι όλη, όλη Τρόικα ελπίζουμε ότι θα παρακολουθήσει το θέμα με επιτυχία και εγώ σου Ουγγαρέζα που έχουμε την Προεδρία μετά, οπότε ήταν ξεκάθαρος ο συντονιστής που μίλησε για το εξάμεινο. Με μεγάλη τους χαρά οι Ευρωπαίοι θα μετέλθουν αυτού του μέσου της πρωτοβουλία. Ήδη είναι στα σκαριά και να δούμε πώς αυτό θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. όπου να είναι θα τεθεί σε ισχύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τον πρόεδρό μας. Σας ευχαριστώ που έγινε η σημερινή συζήτηση. Δεν μπορέσε ο πρόεδρος μας να παραστεί σήμερα, αλλά να ξέρετε ότι είναι στρατευμένος στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λεμασού έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Σεύκοβιτ που μου δίνετε το λόγο πρώτα. Ε, ευχαριστώ του συναδέλφου για τι ε, συστάσει ε, για του εισηγητέ, για τι γνωμοτήσεις των άλλων επιτροπών. Ε, κάποια σχόλια και κάποιε απαντήσει στι ερωτήσει και παρατηρήσει των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Η αρχή την οποία θέλουμε να σεβαστούμε είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτά για τις υπογραφές. Και επομένως το ίδιο συμπεραίνουμε και για τους διοργανωτές που ανήκουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε πολύ αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ή όχι στην Οργανωτική Επιτροπή. Ούτως ή άλλως είμαστε 751 ευρωβουλευτές και χρειάζονται ένα εκατομμύριο υπογραφές. Ας είμαστε λοιπόν ταπεινόφρονες, έτσι. Φυσικά η οχι στην οργανωτικη επιτροπη ουτω η αλλω ειμαστε 751 ευρωβουλευτέ και χρειαζονται ενα εκατομμυριο υπογραφέ. Α ειμαστε λοιπον ταπεινόφρονε, ετσι φυσικα η δικη μα υπογραφή είναι πάρα πολύ σημαντική ποιοτικά, αλλά ποσοτικά δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μία υπογραφή, έτσι. Ο κύριο Ταρκόφσκι Νομίζω ότι μίλησε πολύ σωστά σε ό,τι αφορά τη δράση μας. Έθεσε τα πράγματα στο σωστό μήκο κύματο. Η τροπολογία 119 είναι αποδεκτή και νομίζω από, τα μεγαλύ... από το μεγαλύτερο αριθμό των ευρωβουλευτών. Ας δούμε ποια είναι η ιεράρχηση. Υπάρχουν οι πολίτες των τρίτων χωρών που ζουν, που διαμένουν στις χώρες μας οι κανονικοί, μη εκλεγμένοι πολίτε. οι Ευρωπαίοι πολίτε που ζουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή ε, νομικά πρόσωπα και ιδίω πολιτικά κόμματα. Τι απαντήσει εμεί προτείνουμε. Οι πολίτε των τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να συμμετάσχουν, δεν το επιτρέπει η συνθήκη. Έτσι. Το είπαν πολλοί από εσά, το υπενθύμησαν. Οι, κανονικοί, οι, καθημερινοί Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί και να υπογράψουν και να είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ έκανε μια σημαντική παρατήρηση. Που θα με αναγκάσει να προτείνω ε, μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 119 που λέει στα εθνικά μας κοινοβούλια έχουμε ε, βουλευτές που ανήκουν σε πολιτικά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, προσοχή. Εδώ. Αντίθετα με αυτό που εγώ είχα προτείνει αρχικά, ίσω θα πρέπει να μπλέξουμε του εθνικού βουλευτέ με του ευρωβουλευτέ. Δεν είναι η ίδια κατηγορία κατά ανάγκη. Έχουμε τα μέλη επίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο συμβασμό προτείνω μέσω τη τροπολογία 119 είναι να πούμε μια και αυτό το δικαίωμα δίνεται στους πολίτες, στους απλούς πολίτες. Μόνο αυτοί οι απλοί πολίτες που δεν είναι ευρωβουλευτές, έτσι, βουλευτές και δι ευρωβουλευτές, μπορεί να είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και να μετρηθούν σε αυτά τα 7 ή 8 ή 9 μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Αν όμως τώρα κάποιοι ευρωβουλευτές θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία από την αρχή, μπορούν να βάλουν το όνομά τους στην Οργανωτική Επιτροπή, αλλά η ψήφος τους δεν, δεν μετράει για να θεωρήσουμε ότι έχουμε τον ελάχιστο αριθμό. Μπορεί να είναι 5-10 ας πούμε ευρωβουλευτές που υποστηρίζουν την όλη προσπάθεια μέσα της Οργανωτικής Επιτροπής. Αλλά προσοχή. Τώρα, για τα νομικά πρόσωπα και τα, πολιτικές, τα πολιτικά κόμματα. Μεταξύ των σοσιαλιστών, ας πούμε, Υπάρχουν πολλοί που θέλουν τα πολιτικά κόμματα να ανήκουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Πολλοί από εσά είπανε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης. Μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Φυσικά, αν το ΕΛΚ ή οι σοσιαλιστές οποιαδήποτε, ε, οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή εθνικό κόμμα θέλει να ενθαρρύνει, θέλει να είναι χορηγός, θέλει να βάλει το λογότυπό του, να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί. Μπορεί να το κάνει. Μπράβο του και μπορεί να το κάνει. Και θα είναι εύκολα τα πολιτικά κόμματα που το επιθυμούν να βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο. Με κάθε υποχρέωση όμως διαφάνειας. Οι διοργανωτέ, αν υποστηρίζονται από πολιτικά κόμματα ε, ή από κάποια επιχείρηση, είναι υποχρεωμένοι να το δημοσιεύσουν αυτό το γεγονός. Μίλησα για τους πολίτες των τρίτων χωρών. Έτσι. Ε, μίλησα με τον Άντριου Νταφ για τη δυνατότητα να προβλέψουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει τροποποίηση τη ε, συνθήκη και οι πολίτε μέσω τη πρωτοβουλία των πολιτών να μπορούν να προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τροποποιήσουν τη συνθήκη. Όχι όμω. Λάθο είναι αυτό. Αυτό το νέο άρθρο τη συνθήκη δεν θέλει κάτι τέτοιο. Και ας με διαψεύσει τον Συμβούλιο, κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι εδώ θα προσκρούσουμε στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα, θα θελήσει να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς από αυτό που είμαστε μέχρι τώρα. Και να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η πρωτοβουλία των πολιτών να καταλήξει σε αλλαγή της συνθήκης. Ο κύριος Νταφ ξέρει ότι αυτό εγώ το είχα επιθυμήσει αρχικά στην τροπολογία που είχα καταθέσει στην, ε, Ευρωπαϊκή Συνέλευση. Να φτάσουμε μέχρι την τροποποίηση της ε, συνθήκης. Αλλά προσέχουν σε μια τρομακτική ε, αντίδραση μέσα στη δική μου πολιτική ομάδα, στη δική μου πολιτική οικογένεια και κάηκα, κυρίες και κύριοι. Δεν, δεν θα γίνω τώρα, θα είμαι και στα χαρακόμματα, δεν θα, είμαι και, θα γίνω και Ζαν Ντάρκ, Ιωάννα της Λορένης. Σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις, έγιναν πολλές ε, παρεμβάσεις. Προς την διακατεύθυνση, συγκλίνουσες. Η Κομισιόν δεν είναι τόσο ενθουσιώδης όσο εμεί. Εμεί θέλουμε να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα στην δημόσια κρόαση. Και γιατί αυτό, γιατί. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή. Να αποφύγει να αισθανθεί υποχρεωμένη, πολιτικά υποχρεωμένη, να δώσει ντύ και καλά νομοθετική συνέχεια σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να οδηγεί ντε και καλά σε μια πλειάδα ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Έχουμε υπερβολικά ποτέ πολλά νομοθετήματα. Το ζητούμενο είναι καλύτερα νομοθετήματα, όχι περισσότερα. Θα πρέπει να δοθούν άλλες συνέχειες, λοιπόν. Να εξασφαλίσουμε, λοιπόν, τη δημόσια κρόση, ναι, αλλά όχι το νομοθέτημα ντε και καλά. Θα πρέπει να βρούμε την καλή διατύπωση λοιπόν για να το επιτρέψουμε αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να κρίνει και να συμμετάσχει. Επίσης, από την άλλη, εμείς είμαστε πιο ικανοί να διοργανώσουμε ακροάσεις από την Επιτροπή. Ίσως ο διαμεσολαβητής ή ο ΚΕ, η ΕΟΚΕ η Επιτροπή των Περιφερειών θα μπορούσαν αυτοί να διοργανώσουν ε, δημόσιες ακροάσεις. Ενδιαφέρον και αυτό. Κύριε Μέσο Σμιτ, μέσω της τροπολογίας σας 144 κάνετε μια ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας. Ακριβώ γι' αυτό λοιπόν, για να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει πολιτική συνέχεια διαφορετική από την νομοθεσία, γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε το δικαίωμα αυτό ή τη δυνατότητα αυτή ε, της ακρόασης. Πολλές τροπολογίες, όπως η 144, αλλά και άλλες, ζητούν παρέμβαση του Κοινοβουλίου αναφέροντας ε, την ε, καθήλυν αρμόδια επιτροπή. Εμείς, ε, εμείς στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων λέμε τη δική μας, ας πούμε. Προτείνουμε τη δική μας. Η Επιτροπή Γυναικών τον εαυτό της κτλ. Αλλά απέναντι στην Κομισιόν υπάρχει το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει η Επιτροπή Α, η Επιτροπή Β ή η Επιτροπή Γ. Από εκεί πέρα είναι θέμα δικού μα εσωτερικού κανονισμού να ορίσουμε την αρμόδια επιτροπή. Ο πρόεδρο μίλησε για την προσφυγή στο ΔΕΚ. Δεν θα επανέλθω. Ο κ. Σταρκόφσκι, όπω και ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου, μίλησαν για τη δυνατότητα του να έχουμε ένα ελάχιστο έναν ελάχιστο αριθμό κρατών μελών και ένα ελάχιστο αριθμό πολιτών. Ε, είπαμε λοιπόν, ε, για να βρούμε το, τη λύση, να παραπέμψουμε στη λύση που έχουμε βρει στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Καλή ιδέα. Την κρατάω, γιατί χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια. Αδιαμφισβήτητα, που τα δεχόμαστε όλοι, λογικά αδιασάλευτα. Τελευταία παρατήρηση, επί της οποίας έκανε και ο πρόεδρος Καζίνη, Κασίνη ένα σχόλιο. Είπε ότι το κείμενό μας προβλέπει και ποινική ευθύνη διοργανωτών αν υπάρξουν ανακοινώσεις ή δημοσιοποίησεις προσωπικών δεδομένων κτλ. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει το Εθνικό Κοινοβούλιο να, παρέμβει, να παρέμβει. Θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία δηλαδή, ε, μέσω εφαρμοστικών μέτρων. Στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε πολύ τον τρόπο που δουλεύει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν, ας πούμε, κάθε τόσο βουλευτικέ εκλογέ, σταματάει να δουλεύει το κοινοβούλιο κτλ. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε τότε να πάρει απόφαση. Γι' αυτό μου έρθει μια θαυμάσια ιδέα, Πρόεδρε. Πονηρή θα έλεγα. Ξέρετε ότι η λέξη πονηρός είναι λίγο αμφίσιμη. Και θετική και αρνητική. Έχει κάτι και το και διαβολικό αλλά και θετικό. Τώρα δεν ξέρω εσεί. τι, τι πιστεύετε για την ιδέα που θα σα πω θα ήθελα να μου επιτρέψετε να την αναφέρω στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Για να δω, μόνο και μόνο για να δω, την αντίδραση. Να δω αν θα πάθει καρδιακό επεισόδιο το Συμβούλιο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε το εξή ότι το, ο κανονισμός θα εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή οι νομικές ε, προϋποθέσεις εφαρμογής υπάρχουν σε εννια κράτη-μέλη σε ένα τρίτο ας πούμε μελών. Θα δούμε ποιο είναι αυτός απαραίτητο αριθμό μελών. Ε, το αργότερο, μετά από τόσους μήνες, έτσι. Ποια είναι η αντίδραση. Το Συμβούλιο διαπάντησε. Καρδιακή προσβολή. Παρ' όλα αυτά, παρ' όλα αυτά γίνεται μια, δημιουργείται μια ευγενή άμυλα, έτσι. Αν ας πούμε καθυστερήσει η Γαλλία, θα γίνουν έξαλλοι Γάλλοι πολίτε. Θα πούν Α, οι Βέλγοι, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί κτλ. Έχουν δυνατότητα. Εμεί όχι. Λοιπόν, με ένα ε, ψήγμα πονηριάς σας διατυπώνω αυτή την ιδέα. Σπλήνουμε εδώ τη συζήτηση για την πρωτοβουλία των πολιτών Ευχαριστώ εκ νέου τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς που είναι ήδη μαζί μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, γιατί ολοκληρώθηκε ένας χρόνος από τη θέση σε ισχύ της ε, Συνδίκης της Λισαβόνας και έγιναν πολλά πράγματα έκτοτε, ε, όπως δείχνει και η συζήτησή μας. Ε, τελειώνουμε το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών και ελπίζουμε μέχρι την Άνοιξη να κλείσουμε και την Σύμβαση για τη Διαφύλαξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα πολλά για την ε, διοργάνωση, για τον τρόπο που λειτουργεί η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά ο Αντιπρόεδρος μπορεί να μας πει πολλά και για αυτό ακόμα, αλλά και κυρίως για τη σχέση της Κομισιόν με τα κράτη-μέλη. Γιατί και χάρη στην πρωτοβουλία του κ. Μπαρόζο έχουν γίνει πολλά για τις σχέσεις Κομισιόν και Ευρωπαϊ... Ε, Ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης, ποια είναι η πρακτική στο Κοινοβούλιο, μας, πώς σας φαίνεται αυτή η πρακτική στο Κοινοβούλιο για να εισάγουμε τροπολογίες στις διαδικασίες ε, που αφορούν νομοθετήματα που απορρίπτουμε. Ακόμα, ποιε είναι οι πρακτικέ ε, για τι τροπολογίε που υποβάλλουμε εμεί ε, σε σημεία που η Κομισιόν δεν τροποποιεί. Ε, ζητώ συγγνώμη κύριε Σεύκοβιτς, αλλά θα φύγω αναγκαστικά τώρα. Ε, θα μείνω περίπου ένα τεταρτάκι, γιατί φεύγει το αεροπλάνο μου για την Αφρική, για την Κινσάσα, όπου θα γίνει η συνεδρίαση των α, χωρών ΑΚΕ. Ε, σας δίνω λοιπόν τώρα το λόγο και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, γιατί θα σας δω μετά στο τέλος. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να συζητήσω με την Επιτροπή συνταγματικών θεμάτων και να συζητήσω για τα θέματα της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρετε ότι ήταν θαυμάσιος ο χρονισμός και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να δούμε το χρόνο ο οποίος διέρευσε και ο οποίος είναι έτοιμος να τελειώσει για το σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Κάποια πράγματα ήταν σχεδόν αυτόματα, από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια νύχτα στην άλλη, είχαμε μια νέα θεσμική δομή. Είπα το εκπρόσωπο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, είχαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου, πράγματα τα οποία θέλαμε πάρα πολύ καιρό, μια ενιαία νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρεμίσαμε και τους πυλώνες. Και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έγινε νομικά δεσμευτική και είδαμε μια σαφή ενίσχυση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορους τομείς και είδαμε επίσης ότι η κοινοτική, η ενωσιακή όπως τη λένε τώρα μέθοδος έχει ε, εδρεωθεί πλήρως στην καθημερινή μας συνεργασία και την καθημερινή μας ζωή. Είδαμε επίσης να υπάρχει και αυξανόμενο ενδιαφέρον και θα επανέλθω στο θέμα αυτό για την νομοθετική δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων που προσπαθούν να δουν πώς θα αυξήσουν τη δική τους συμμετοχή θέλουν να μελετήσουν τη διαδικασία αυτή και να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όλα αυτά είναι αλλαγές λοιπόν οι οποίες επεσυνέβησαν που ήταν από κύμα της αυτόματης κατά κάποιο τρόπο θέσης εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά που έπρεπε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, διότι ήταν επιταγέ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Παραδείγματο χάρη το θέμα τη ε, νομική, ε, την τροποποίηση νομικής, νομικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέματα όπως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής δράση Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν εάν δεν υπήρχε αυτό το θαυμάσιο συνεργατικό πνεύμα μεταξύ της Κομισιόν και της Επιτροπής σας και ευρύτερα μεταξύ της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω να τα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου για να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα συνεργασίες, γιατί έχω κάθε ελπίδα ότι θα εγκριθεί μέσα στο Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και θα μπορέσουμε να έχουμε και την απαραίτητη πρόοδο για τα θέματα των εφαρμοστικών και κατεχώρηση πράξεων. Θέλω σα σας ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε για το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο διευθύνεται αυτή την Επιτροπή και επιτρέπετε στην Κομισιόν να είναι πάντα παρούσα στις συνεδριάσεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντονιστές του συζητητέ για, για, αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα θέματα, γιατί χωρί τη συνεργασία του δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τα πάρα πολύ στενά χρονοδιαγράμματα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Εμεί εισάγουμε το νέο νομικό πλαίσιο σε δύσκολες στιγμές. Ήδη στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του αυτό το πλαίσιο δοκιμάστηκε ιδιαίτερα γιατί δεν έχουμε δει ποτέ τόσο μεγάλη οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είδαμε ποτέ τόσο δύσκολη δημοσιονομική ε, κατάσταση και χρειάστηκε να συνδυάσουμε αυτή την κρίση με το νέο νομικό πλαίσιο. Το γεγονό ότι βρήκαμε καλέ λύσει, όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν σωστή η συνδίκη τη Λισαβόνα, ότι λειτουργεί το πλαίσιο τη Λισαβόνα και απλώ χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κάτι για τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπω προτείνατε και εσεί να πω στην πρόσκλησή σα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια ήδη από το 2006 όταν ξεκινήσαμε τον πολιτικό διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν οποιαδήποτε πρόταση ή πρωτοβουλία της Κομισιόν. the... Και λειτουργεί αυτό μέχρι σήμερα. Αλλά με την, με την θέση εφαρμογής της Συνδίκης Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό... τα Κοινοβούλια έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα βάσει του πρωτοκόλου 2 και της διατότητα επικουρικότητα να προσφέρουν τι προτάσει του επί οποιασδήποτε νομοθετικής ε, πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε πάρει πάνω από 150 απόψεις από τα, Ευρω... από τα Εθνικά Κοινοβούλια για νομοθετήματα της Κομισιόν. Και αν συνδυάσω τον πολιτικό διάλογο και τη διαδικασία επικουρικότητας, πάνω από 250 συνεισφορές έχουμε λάβει από το Φεβρουάριο του 2009, 2010 συγγνώμη. Και είχαμε πάνω από 150 γνώμες από τα Εθνικά Κοινοβούλια όταν από του, από το ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος. Μόνο 24 εκ των οποίων ήταν ε, αρνητικές και επομένως ούτε η κίτρινη ούτε η κόκκινη κάρτα έχουν ακόμα ε, επιδειχθεί από τα κράτη-μέλη από τα κοινοβούλια μάλλον. Ε, είχαμε δύο προτάσεις κομισιών, μία για τους εποχιακά εργαζόμενους και η άλλη ήταν για τις εγγύησεις των καταθέσεων, οι οποίες έτυχαν αρνητικών γνωμοδοτήσεων. Προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των κρατών και θα τους δώσουμε τις απαντήσεις μας όσον νούπο. Επίσης για τους εποχιακά εργαζομένους είχαμε ίσο αριθμό θετικών και αρνητικών απόψεων. Νομίζω λοιπόν ήταν ισορροπημένη η προσέγγισή μας. Είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε μια τέτοια έντονη διαφοροποίηση απόψεων και θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τις απαντήσεις μας στις γνωμοδοτήσεις αυτές των Εθνικών Κοινοβουλίων πάρα πολύ προσεκτικά. Πώς λοιπόν λειτουργεί ο μηχανισμός ελέγχου της επικουρικότητος, όπως όλα τα νέα συστήματα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως. Οι περισσότερε γνωμοδοτήσει έρχονται από τι γερουσίε, τι άνω όπου υπάρχει περισσότερο χρόνο, και από τα κοινοβούλια που έχουν ήδη θεσπίσει δίκτυα εμπειρογνωμόνων για να υποστηρίζουν τι επιτροπέ οι οποίε ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ε, τεκτενόμενα. Βλέπουμε όμω να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα τα κοινοβούλια που θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο και στον πολιτικό διάλογο και στο μηχανισμό ελέγχου της επικουρικότητος για την ε, επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την Επιτροπή. Γιατί η Κομισιόν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω την επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί ατενίζουμε τα κοινοβούλια αυτά ως σημαντικούς συμμάχους σε πολλούς τομείς. Παραδείγματο χάρη η Ευρώπη 2020. Θέλουμε συμμετοχή όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θέλουμε να εμπλέξουμε τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια σε μεγαλύτερη συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις για να μπορέσουν να ε, εκπονηθούν τα καλύτερα προγράμματα μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο για να υποστηρίξουν την Ευρώπη του 2020. Χωρίς τέτοια προγράμματα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνορο. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλα τα θέματα του προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε θέλουμε να ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ήδη από τα μέσα του Ιανουαρίου 2011 ώστε να γίνει η αξιολόγηση από την Κομισιόν και μετά από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ για το κατά πόσο οι προτινόμενες παράμετροι για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και ελληνικά σχέδια τηρούν το κριτήριο της αηφορίας και βιωσιμότητας. Έτσι λοιπόν, αν τα εθνικά κοινοβούλια έχουν όλη αυτή την πληροφορία, θα μπορούν να πιέζουν τι κυβερνήσεις του για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των σχεδίων αυτών και θα έχουν μια προσθέμενη αξία οι συζητήσει για τα θέματα αυτά. Θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία για τα εθνικά κοινοβούλια για καλύτερη μεταγραφή και μεταφορά του ευρωπαϊκού δικτύου, δικαίου. Είχα μια τέτοια συζήτηση την Πέμπτη και θεωρούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα είναι οι σύμμαχοί μας για να μην υπάρχουν πρόσθετες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όταν μεταφέρεται στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Και βλέπουμε, βλέπετε και εσείς πόσο δύσκολο είναι το θέμα του προπολογισμού για το 2011 και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο θα είναι συζήτηση και για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο, αυτό το διάβολο επικοινωνία για να συζητήσουμε και τι απόψει μα και με τα Εθνικά Κοινοβουλία αυτό το προπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι με τη χρήση αυτών των διάβλων επικοινωνία και με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία και τι Ευρωπαϊκέ Συζητήσει θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα ευρωπαϊκά θέματα και στο τοπικό επίπεδο εθνικό επίπεδο. Θα συζητείται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εθνικά κοινοβούλια και έτσι δεν θα έχουμε εκλογέ οι οποίε γίνονται ευρωεκλογέ μονάχα επί τη βάση εθνικών θεμάτων. Και πιστεύουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει την Κομισιόν να αναπτύξει περισσότερο τη σχέση τη με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί ήδη υπάρχει μια συνεργασία που έχει προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε ήδη στι εισαγωγικέ σα παρατηρήσεις σε προτάσεις αναδιατύπωσης νομοθετημάτων. Η διαδικασία αυτή η αναδιατύπωση είχε σαν στόχο να διευκολύνει τη ζωή μας. Αν έχετε νομοθεσία η οποία χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, η Κομισιόν μπορεί να υποβάλει προτάσεις τροποποίησεως αυτής της νομοθεσίας και εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτές τις τροπολογίες. Είδαμε λοιπόν έναν τρόπο να υλοποιήσουμε το δικαίωμα Πρωτοβουλίε τη Κομισιόν παράλληλα επιταχύνοντα το νομοθετικό έργο χωρί να χρησιμοποιούμε την πλήρη διαδικασία για μια αλλαγή της νομοθεσίας η οποία θα μπορούσε να είναι στο μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσία ακόμα θετική και απλώς μερικές λεπτομέρειες έπρεπε να αλλάξουν. Και επιζητήσαμε να έχουμε τις απόψεις και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία αναδιατύπωσης και αν θα έπρεπε υπήρξε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μεταξύ Προέδρου Μπαρός και Προέδρου ε, Μπούζεκ και είναι σημαντικό να επανέλθουμε στη συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, των βασικών θεσμικών οργάνων για την καλύτερη ε, συνεργασία και την καλύτερη χρήση της διαδικασίας αναθεώρηση αναθεώρησης για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιτάχυνση της νομοθετικής εργασίας μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στα θέματα της πρωτοβουλίας πολιτών, γιατί άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ε, είπε και ο κύριος Λαμασούρ και η κυρία Γκουρμάη και ήταν πολύ ε, δημιουργική και πολύ καλή η ατμόσφαιρα εδώ. Όταν πηγαίνει κανεί σε ένα τριγωνικό διάλογο, πολλέ φορέ περιμένει πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει. Με του εισηγητέ σα όμω είναι πάντα διασκεδαστικό, έχει πάντα ενδιαφέρον και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Τώρα, τι σημαίνει καλή συμφωνία από την πλευρά τη Κομισιόν. Ξέρετε ότι εμεί πιστεύουμε ότι οι ακρόασει θα πρέπει να οργανώνονται πάντα από το Κοινοβούλιο με τη βοήθεια της Κομισιόν για τους συγκεκριμένους λόγους που ανέφερε ο Αλέν Λαμασούρ. Η Κομισιόν πρέπει να δώσει την τελική ανακοίνωση για το πώς πρέπει να δοθεί συνέχεια σε μια πρωτοβουλία πολιτών, γι' αυτό πρέπει να είναι κάπως αποχωρισμένη από τη διαδικασία που εκτιλήσεται μεταξύ της ε, τελικής απόλυξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών και της απάντησης που δίνεται από την Κομισιόν είχαμε πολλές συζητήσεις για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θέλω να κάνω σαφές για την υποστήριξη που πρέπει να δίνει η Κομισιόν. Τονίσαμε ότι εμείς θέλουμε να υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν μια πρωτοβουλία πολιτών και θα έχουμε και μια δήλωση για το πώς θα γίνεται αυτή η βοήθεια, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να τεθεί μέσα στο κείμενο της νομοθεσίας γιατί αυτό μπορεί να βγει σε νομικές αντιπαραθέσεις, ανεπαρκές, τι ακριβώς σημαίνει, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαμαχών. Γι' αυτό προτιμούμε επίσης να υπάρχει και μία μονάχα ενιαία λογή, γλωσσική μορφή όταν έχουμε <clears throat> να κάνουμε τη διαδικασία καταγραφής, έτσι είμαστε πάρα πολύ σαφείς για το τι ακριβώς καταγράφει. Αν θέλουν να προσθέσουν στη συνέχεια άλλες γλωσσικές μορφές οι οργανωτές, είμαστε πάντα έτοιμοι να το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι να δούμε αν υπάρχουν και αντιφάσεις μεταξύ των γλωσσικών μορφών. Και κάτι το οποίο είναι προσφυλές στην κυρία Γκουρμάη, πώς θα πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση στο μέλλον, η επανεξέταση αν θέλετε, για την διαδικασία. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά χωρίς να έχουμε μια τόσο λεπτομερή, τόσο λεπτομερής προδιαγραφές, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση ότι ήδη τώρα που εγκρίνουμε το νομοθέτημα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να το δοκιμάσουμε πρώτα, να δούμε πώ λειτουργεί και μετά μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εν ευθέτω χρόνο να τροποποιήσουμε το νομοθέτημα αυτό. Και φυσικά αν έχουμε ένα κεντρικό, μια κεντρική ιστοσελίδα θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα γιατί μπορούμε έτσι να έχουμε ένα κοινό λογισμικό για όλους τους οργανωτές. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και την Αντιπρόεδρο κυρία Βόλις γιατί νομίζω μπορέσαμε να πετύχουμε πολλά πράγματα για το μητρό διαφάνειες γιατί αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει πιο διάφανος έλεγχος της νομοθετικής διαδικασίας της Βρυξέλλες. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπογραφεί αυτό εν συντομία και νομίζω και το Συμβούλιο η Βελική Προεδρία έπαιξε σημαντικό ρόλο και η Ουγγρική Προεδρία έχει τονίσει ότι της ενδιαφέρει να συνεχίσει. Επίσης το θέμα των πινάκων συσχετισμού που συζητήθηκε την Πέμπτη, εγώ είμαι ιδιαίτερα υπόχρεος στον πρόεδρο Μπούζεκ και στη συνέλευση των προέδρων των πολιτικών ομάδων που προσπαθούν να δουν τρόπους με τους οποίους οι πίνακες συσχετισμού μπορούν να είναι τμήματα της νομοθεσίας γιατί εξασφαλίζει και τη σωστή εφαρμογή στα κρατη τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την κάνει πιο επακρίβη. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν δύσκολο το έργο σα σε πολύ δύσκολε συνθήκε, αλλά τα εγχειρήματα στα οποία αποδεθήκαμε από κοινού ήταν πράγματι πολύ επιτυχή μέσα στον πρώτο χρόνο που λειτουργούμε στο, πρώτο, στο πλαίσιο αυτό της Λισαβόνα ε, Λισαβόνας και προσβλέπω και σε περαιτέρω συνεργασία στο τέλος του χρόνου και του χρόνου επίση. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Όπως σας είχα πει και πριν, ε, πρέπει να φύγω τώρα. Ε, θα δώσω το, τη θέση του Προέδρου στην κυρία Γκουρμάη για να ακολουθήσει συζήτηση πάνω στην ε, παρέμβασή σας. So, dear uh, Commissioner... Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η χρονιά. Είχαμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ε, το πλαίσιο το έθεσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, χαίρομαι που έχετε ενθουσιασμό, δέσμευση. Το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Η γραμματεία που ετοίμασε την συνεδρίαση έβαλε το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών όχι τυχαία στη μερίσια διάταξη. Γιατί θέλαμε να ακούσετε και εσείς προσωπικά. Ε, έχετε μια θαυμάσια ομάδα που σας περιβάλλει και που σας προετοιμάζει και εγώ ως ε, μέλος ε, του ανεπίσημου τρίου αυτού. Συμμετείχα στις ε, συζητήσεις. Δεν θα αντιδράσω στα όσα είπατε, γιατί πρέπει να γίνει μια συζήτηση τώρα. Ο κύριος Γκερέρο έχει τον λόγο πρώτος και μετά ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που παρίσταστε σε αυτή τη συνεδρίαση. Η παρουσία σας στην Επιτροπή μας είναι συχνή και τα μέλη της Επιτροπής ε, σας είμαστε ευγνώμονες για αυτή την ε, δέσμευσή σας. Είπατε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είχε δύο μεγάλα πακέτα μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Η πατή εκπρόσωπος, ο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και από την άλλη μεταρρυθμίσεις που είχα σαν σκοπό να ενσωματώσουμε τους πολίτες στον, στην ε, ευρωπαϊκή οικοδόμηση και τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα είναι πολύ πιο συμμετοχικό και θα εντάξει και τον πολίτη και τους εθνικούς βουλευτές των 27 κρατών μελών στη διαδικασία λειτουργίας. Για αυτή την περίπλοκη διαδικασία. Και σήμερα <laughs> δηλαδή Ακριβώς γι' αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι μπορέσαμε να το συζητήσουμε δύο φορές εδώ. Πρώτα-πρώτα από τους τη ε, της Επιτροπή και τώρα από τον υψηλό τη εκπρόσωπο. Οπότε και εγώ οφείλω να σας πω ότι ε, δεν είχα καμία αντίρρηση, συνέπεσαν οι απόψει μας και την πρώτη φορά που το άκουσα και τη δεύτερη. Αλλά αυτό πάντοτε είναι πάρα πολύ θετικό να το ακούει κανένα από κάποιον υψηλά ιστάμινο. Τον το... Γιατί αυτό σημαίνει δέσμευση. Πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή για τα εθνικά κοινοβούλια. Πάρα πολύ σωστό είναι να, να ακούγεται η γνώμη του Επιτρόπου, διότι πάρα πολύ συχνά τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να χωνέψουν ακριβώς τι τους ζητείτε, τι τους ζητείτε σε σχέση με τη συμβολή τους ή στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, διότι σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια υπάρχει ένα επίπεδο, ένας βαθμός εσωτερικής ε, σύγκρουσης. Σε όλες τις χώρες πολύ συχνά θεωρούν ότι δεν είναι θέμα προτεραιότητας το να δεσμευθούν όσον αφορά ε, το τι γίνεται με τα ζητήματα τα οποία τώρα ε, είναι επίκαιρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είναι και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό το ότι συχνά οι πρόεδροι των ε, εθνικών κοινοβουλίων έχουν κάποιου δεσμεύσει εθνικές και συνήθως στέλνουν τι συναντήσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δυστυχώς, όποιον ευκαιρεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό μας οδηγεί στο να έρχεται κάθε φορά διαφορετικός και αφού είναι διαφορετικός δεν είναι δυνατόν κανείς να ξέρει τι έγινε, να υπάρχει κάποια συνέχεια, να υπάρχει κάποιο είδους ε, συμμετοχή, δέσμευση προσωπική για τις εργασίες αυτές. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, μου άρεσε κάτι σχετικό το οποίο είπε ο Επίτροπος, που, γιατί έτσι είναι δυνατόν να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς την επίλυση του σχετικού προβλήματος. Δηλαδή να γίνουν πιο στενές οι σχέσεις με τις αντίστοιχες επιτροπές τις κοινοβουλευτικές των εθνικών κοινοβουλίων εκείνες οι οποίες έχουν την ανάλογη αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων και ας πούμε στην περίπτωση της Ισπανίας, έχουμε άνω και κάτω βουλή, έχουμε βουλευτές και γερουσιαστάς και έχουμε μια μεικτή επιτροπή για τις ευρωπαϊκέ υποθέσεις όπου συμμετέχουν και βουλευτές και γερουσιαστές. Ε, Βεβαίω και είναι δυσχερές να μπορέσουμε αυτή η ε, μεικτή επιτροπή να πούμε ότι αναλαμβάνει την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου μας. Αλλά η στενή συνεργασία με αυτή τη μικρή επιτροπή τότε αυτή πρόκειται να διαβιβάσει το σχετικό μήνυμα στο κοινοβουλίο μας. Και αυτό θέλω να σας προτείνω. Έχουμε άλλωστε και τον κύριο Μέντε που έχει την απαραίτητη εμπειρία και ταυτίζονται οι του σε αυτό το σημείο με τη δική μου. Είναι το να μπορέσουμε να ε, βρούμε μια πλατφόρμα σταθερή συνάντησης Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων και να δούμε ποια είναι η ομόλογη επιτροπή μας, αυτή η οποία ασχολείται με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, να πρόκειται για έναν μηχανισμό διαμεσολάβησης μεταξύ ημών εδώ και εκείνων. Και αυτό να γίνεται έστω και με άτυπο τρόπο να εμπλέκονται όλο ένα και περισσότερο σε αυτά τα θέματα μας τα εθνικά κοινοβούλια και με το, το πέρασμα του χρόνου κατά κάποιο τρόπο πρόκειται να ε, διαπιστωθεί ακριβώς πώς γίνεται η διαδικασία λήψη αποφάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, το δικό μας, αυτά τα οποία και εκεί συζητούν στο δικό τους, το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται να έχουμε ε, περισσότερη συνέργεια, πιο στενές σχέσεις. Πάντως, τη σημερινή μέρα βρισκόμαστε σε κάποιο είδους ε, αποτελμάτωση, σε κάποιο είδους ε, ανησυχία και ένταση και στρες. Τι γίνεται με την οικονομία, τι γίνεται με το ευρώ, τι γίνεται με την απάντηση που πρέπει να δώσουν τα ευρωπαϊκά όργανα σε αυτά τα προβλήματα για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει επομένω να καταλάβουν τα εθνικά κοινοβούλια το ότι η, η πτυχή ευρωπαϊκή είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ερίκε, ο Ανδρέας Νταφ. Και μετά ο Ινίγο με Μέντες Δεβίβο. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Εάν όχι, κλείνω τον κατάλογο. Εγώ συμφωνώ πραγματικά με αυτά που ελέγχθηκαν ότι μέχρι στιγμή η συζήτηση της έχει εφαρμοστεί πολύ καλά, αποτελεσματικά, αποδοτικά και από την Κομισιό και το Κοινοβούλιο. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για το αν μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επενετικές παρατηρήσεις και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να διανεμηθεί και πάλι στα μέλη του Συμβουλίου, μήπως και τη διαβάσουν ίσως να την καταλάβουν πληρέστερα από ό,τι φαίνεται να την έχουν κατανοήσει μέχρι στιγμής. Βέβαια, βρισκόμαστε και πάλι στην φάση που θα πρέπει να αλλάξουν και πάλι οι συνθήκες. Είμαστε σε μια τέτοια φάση λοιπόν και η συνεργασία μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι ουσιαστική. Θα πρέπει να αλλάξει αλλάξει το οικονομικό σύστημα. Για να υπάρχει ένα σταθερό σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα ενδεχόμενης ε, αδυναμίας εξυπηρέτησης του κυριαρχού του χρέους κυριαρχών κρατών. Και αυτό είναι ένα τμήμα του μηχανισμού. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή γιατί σημαίνει στην πράξη ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί να βρίσκεται σε μια φάση μόνιμης κρίσης. Μέχρι στιγμής έχει υπάρξει ένα πλαίσιο βάσει του άρθρου 122 που είναι το άρθρο το οποίο καλύπτει εθνικές καταστροφές, φυσικές καταστροφές εκτάκτου χαρακτήρα πέραν της δύναμης αντιμετωπίσεως των εθνικών κρατών. Όσο το σκεφτόμαστε περισσότερο αυτό, βλέπουμε ότι το άρθρο 122 δεν είναι ακριβώς <clears throat> η καταλληλότερη νομική βάση για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους μηχανισμών κρίσης, για την αντιμετώπιση κρίσεων οικονομικών όπως αυτές που βλέπουμε τώρα και γι' αυτό βλέπουμε και το άρθρο 136 το οποίο αφορά ειδικότερα και προς το παρόν αποκλειστικά τη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνη η Κομισιόν τώρα ότι το άρθρο 136 είναι πιο κατάλληλο άρθρο, μια καταλληλότερη νομική βάση για ένα τέτοιο μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων από το άρθρο 122. Εάν ούτω σκέφτεται η Κομισιόν, τι θα πράξετε για να συνδέσετε και τα κράτη που αυτή τη στιγμή είναι εκτός του ενιαίου νομίσματος, όπως η Πολωνία και η Σουηδία, ε, αλλά και χώρες οι οποίες είναι με πρόθεση να μπουν στη ζώνη του ευρώ μόλις μπορέσουν, μόλις εκπληρώσουν τα απαραίτητα κριτήρια σύγκλησης. Κράτη δηλαδή που έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι είναι απόλυτα έτοιμα να συνεργαστούν για την οικοδόμηση του μηχανισμού αυτού ο οποίος προβλέπεται. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη του κυρίου Επιτρόπου για την νομική βάση. Δεύτερον, θεωρείτε μήπως ότι μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στη δομή και στη λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να τύχει συμφωνίες μέσα στο μηχανισμό, μέσα στον απλοποιημένο μηχανισμό αναθεώρησης της ε, συνθήκης βάσει άρθρου 48 παράγραφος 6. Εάν υπάρξει μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να είμαστε ε, σίγουροι ότι δεν υπάρχει αύξηση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βλέπω το θέμα αυτό υπό το πρίσμα της ακαδημαϊκής και αντιπαραθετικής κατά κάποιο τρόπο συζήτησης που, περιλα... που πε... περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα και αναρωτιέμαι πράγματι αν η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων αν πράγματι δεν αυξάνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τις επεκτείνει. Και δεν είναι μονάχα αυτό ένα θέμα πολιτικής επιλογής. Αυτό θα πρέπει να έχει και απόλυτη νομική σαφήνεια για να μας προστατεύσει από διαμφισβητήσεις και προσφυγές στα δικαστήρια κατά της νέας συνθήκης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις τουλάχιστον της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Τέλος, πιστεύω θα έχετε δει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δημοσίευσει ένα νομοθέτημα που έχει σαν στόχο να αλλάξει τους όρους της Βρετανικής συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το να προτείνονται ε, δημοψηφίσματα σε όλες τις ε, σημαντικές αλλαγές της συνθήκες και για τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων διατάξεων πασαρέλας που περιλαμβάνει η συνθήκη και επίσης σε σχέση με το μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Εάν η Μεγάλη Βρετανία, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο καλύτερα, μπει σε αυτή την ομάδα η οποία συμμετέχει σε μια διαδικασία ε, συνεργασίας. Αυτό είναι ίσως ένα απομακρυσμένο σενάριο, αλλά ούτως ή άλλως είναι ενδεχόμενο να υπάρξει ευρύτερη χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι το οποίο κατά την απόψή μου μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση του θεσμικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως θα θα φέρει τους Βρετανούς υπουργούς σε αντιπαράθεση με τις διατάξεις της συνθήκης που τους υποχρεώνει να δεσμεύουν με αυτά που αποφασίζουν στο Συμβούλιο Υπουργών της κυβέρνησης τους. Είναι το άρθρο 16.2. Υποχρεώνει τους υπουργούς να είναι σε θέση να δεσμεύσουν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους κόλπους του Συμβουλίου. Αν μετά όμως από μία απόφαση στο Συμβούλιο θα πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα για ηλιμένες αποφάσεις, αυτό σίγουρα θέτει προβλήματα για την ε, νομιμοποίηση της Βρετανικής συμμετοχής στο Συμβούλιο των Υπουργών. Δεν περιμένω η Κομισιόν να έχει ήδη αξιολογήσει πλήρως την ε, σημασία και τις επιπτώσεις αυτού του νομοθετήματος, αλλά σας το επισημαίνω ως ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να τύχει συζήτηση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάθε λόγο και νομιμοποιείται να εκφράζει την, ε, ε, την ανησυχία του για αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, μετά από όλα αυτά τους πετάξετε έξω έξω μετά από όσο είπε ο κ. Νταφ, έξω από το Συμβούλιο. Εγώ όμω, οποία χαρά σα, θα είμαι πολύ πιο φιλικό και άκουσα όσα μα είπατε, κύριε Επίτροπε, στην εισήγησή σα για την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων ει τα τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αυτό το σύστημα τη έγκαιρη προειδοποίηση, το οποίο και εθεσπίσαμε Οπότε και θεσπίστηκε αυτή η διαδικασία με τις κάρτες όταν η πλειοψηφία των ε, κοινοβουλίων έχει κάποιες θεμητές αμφιβολίες και επιφυλάξεις για την ε, επικουρικότητα. Όχι την αναλογικότητα, την επικουρικότητα λέγω και ανέκαθεν εγώ επρέσβευα ότι αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Στην πράξη πάντως τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι σαν αναμέτρηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ανέκαθεν έλεγα και το είχα πει ότι στην πράξη έχουν πάρα πολλέ χώρε που θα μπορούσαν να έχουν την ίδια άποψη, οπότε γι' αυτό την ενδυναμώνει την άποψη αυτή. Αλλά αν έχουμε ένα μόνο. Οι δυο κοινοβούλια τα οποία διατηρούν κάποιε θεμητέ επιφυλάξει. Ε, αυτό δεν είπα να πει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη και αυτό ισχύει και για μα. Και για μα ε, ότι θα πρέπει και εμεί να το λάβουμε υπόψη και αυτό να περιληφθεί στι δικέ μα θέσει. Ε, όσον αφορά δε δύο σχέδια νομοθετημάτων, να έχουμε κάποιες απόψεις των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε. Αυτό έχει σημασία, σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Και αυτό όχι σαν μια στοιχειώδης ευγένεια, σαν πρωτόκολλο γεωρευτικό, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σχέσεις σχέση ημών και εκείνων. Επομένω, η ανταπόκριση, η απάντηση, η απόκριση έχει μεγάλη σημασία αυτό να σου πω. Επίσης, με την ευκαιρία, Πρόεδρε, που έχετε τέτοια αρμοδιότητα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και κυρία Πρόεδρε, έτσι, προκαταλαμβάνω αυτό το οποίο θα κουβεντιάσουμε ίσως εδώ, για να δούμε, να ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν όσον αφορά την έγκριση του προπολογισμού για τη χρήση του 11. Και σας λέω έτσι την προσωπική μου άποψη. Όμως τη σημερινή μέρα που η Ευρώπη μαστίζεται από αυτή τη σοβαρή και βαθιά κρίση θεωρώ ότι το να μην έχει προϋπολογισμό ένωση για το 2011 είναι το λάθος πολιτικό μήνυμα. Καταλαβαίνουμε τους λόγους, αλλά πολλοί δεν τους καταλαβαίνουν και πιστεύουν ότι αυτό το οποίο σήμερα θα πρέπει να γίνει είναι ο ένας να στρίξει τον άλλο, να τον βοηθήσει τι να, να πάμε σε αυτή την παράδοξη, την περίεργη λύση των τιμωρίων, Αυτό δυσκολεύει τη ζωή των κρατών μελών. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Νομίζω ότι κάπως άλλες τα πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο. Κύριε Αντιπρόεδρε, πέστε μας, τι πρεσβεύετε, τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Να ξέρετε ότι πάντοτε σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον και πάντοτε είναι ευχάριστη η παρουσία σας εδώ. for um, Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Και τώρα είναι ίνκη και η μεγάλη στιγμή να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο. να υπενθυμίσω όμως ότι μια και συναντώμεθα τακτικά, καλό θα ήταν να σκεφτούμε ποιο θα ήταν η επόμενη συνάντησή μας και το θέμα το οποίο θα θέλαμε να ακούσουμε από τον Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Ενρίκε Γερέρο. Τα εθνικά κοινοβούλια γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν αυτό το νέο εργαλείο, ε, με το οποίο μπορούν ε, να έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπάρχει μια αναζήτηση στα ευρωπαϊκά, στα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά αυτό το εργαλείο. Όταν τους επισκέπτομαι, μου λένε ότι οι οχτώ εβδομάδες που ε, μας δίδεται για να αντιδράσουμε δεν είναι αρκετά μεγάλο διάστημα για να αντιδράσουμε σε όλες τις προτάσεις. Η απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα είναι συνήθως ότι είναι πολύ σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να θεσπίσουν τις δικές τους προτεραιότητες. Φαντάζομαι ότι για την Ισπανία οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση για την αλληλεία είναι πολύ σημαντική, ενώ για τη χώρα μου, ας πούμε, τη Σλοβακία, δεν είναι πολύ σημαντικές προτάσεις αυτές. Και επομένως ε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια και το κοινό πραγματικά εκ των προτέρων για το πρόγραμμα εργασία της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τις επερχόμενες χρονιές, ούτως ώστε να βλέπουν την ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορούν να εστιάζουν την προσοχή του ε, και την ενέργειά του, βέβαια εκεί που του ενδιαφέρει περισσότερο. Είναι πολύ πρακτικό τρόπο αυτό και πολύ συνετό και βλέπω ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτόν τον τρόπο εργασία. Είχα την ε, ευκαιρία με τον να συζητήσω με τον κύριο Αρία Κανέτα, τον ε, πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής στην Ισπανία, ε, και ακριβώς αυτή η αντίδραση, την αντίδραση άκουσα και από αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό να ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας. Αυτό είπε. Και είπε επίση ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλό θα ήταν να είναι σε πιο συχνή επαφή με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, συχνά ακούμε διαφορετικές απόψεις Δηλαδή, βουλευτές από το ίδιο κόμμα, ε, εθνική και ευρωπαϊκή, εκφράζουν διαφορετικές θέσεις. Ε, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πραγματική επικοινωνία. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη επαφή. Ε, να υπάρχει ένα σημείο το οποίο λαμβάνει την πληροφορία από την Επιτροπή και μετά την διαχέει. Αυτό το, το πράγμα προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε ακόμα, αυτό το σημείο επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και να στέλνουμε δηλαδή όλε μα τι πληροφορίε εμεί και από το σημείο αυτό επαφής θα λαμβάνουμε την επιβεβαίωση ότι όντως ελήφθησαν οι προτάσεις ή δεν ελήφθησαν αντίστοιχα για το νομοθετικό μας έργο. Ακόμα πιο σημαντικό για τα εθνικά κοινοβούλια στο μέλλον θα είναι το να αποφασίζουν οι ποια είναι τα θέματα, ποιοι είναι οι φάκελοι που θα αποφασίζονται από τη μεικτή επιτροπή ή αν θα πρέπει ας πούμε, να έχουμε εξειδικευμένε επιτροπέ, φερειπίνα γεωργικά θέματα. Ή να συμμετέχει σε αυτή τη μεικτή επιτροπή και ε, ειδική επιτροπή για τα γεωργικά θέματα. Και να πηγαίνει μάλιστα και ο, ο Υπουργός ο οποίο συμμετέχει στα συμβούλια σε αυτές τις μικτές επιτροπές, ούτω ώστε να εμπλακούν περισσότερο στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Τέλος. Η προσωπική μου γνώμη για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές επαφές, υπάρχει κόζακα, Ξέρετε πολύ καλά ότι τα άτομα έρχονται και παρέρχονται. Επομένως, δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει μια μόνιμη ας πούμε, σχέση με την Ευρώπη. Ελπίζουμε λοιπόν αυτός ο νέος μηχανισμός με τις μεικτές επιτροπές θα οδηγήσει σε μια εξειδίκευση, αν θέλετε, για τα ευρωπαϊκά θέματα στα, ευρωπαϊκά, στα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή να, έχει ένα, να υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό που θα, ε, που θα ασχολείται συνέχεια με τα ευρωπαϊκά θέματα και ο καθένας να γνωρίζει με ποια ευρωπαϊκή συγκεκριμένα επιτροπή ασχολείται κτλ. Ο κύριο Νταφ ε, δεν είναι μόνο ευρωβουλευτή, αλλά είναι και λόγιο. Όταν μου κάνει ερωτήσει, πάντα λοιπόν ε, λούζω με κρύο υδρότα αλλά αυτή τη φορά με προειδοποίησε. Ήταν τόσο ευγενικό. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησα να μελετήσω και να έρθω ε, έτοιμος, αλλά δεν ξέρω αν θα τον ικανοποιήσω παρόλα αυτά. Για την αλλαγή της συνθήκης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, κύριε Νταφ, ε, συζητούσαμε για τη συνθήκη. Δεν θα φανταζόσασταν ένα χρόνο πριν ότι ένα χρόνο μετά θα συζητούσαμε ξανά για αλλαγή τη συνθήκη. Πάντω τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, έγινε αυτό το τεράστιο έργο. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν να διερευνήσουμε όλες τις πιθανές νομικές οδούς και ατραπούς για να βρούμε τη λύση στη δημιουργία αυτού του νέου μόνιμου μηχανισμού στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου και των ευρωπαϊκών συνθήκων. Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε δίνοντας ε, εντολή στο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναζητήσει και να διερευνήσει τις απόψεις των κρατών μελών, ούτω ώστε να ετοιμαστούν οι λύσεις για πιθανή αλλαγή των συνθήκων. Από χθε έχουμε καλά νέα. Οι Υπουργοί των Οικονομικών ε, καταλήγουν στις προτάσεις τους για αυτό το μηχανισμό που θα είναι, ελπίζουμε, έτοιμος το 2013. Θα είναι πολύ πιο έτοιμος, ε, έτοιμος να λειτουργήσει, θα εμπλέξει πολύ περισσότερο τον, τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που έλειπε από τους τρέχοντες μηχανισμούς και από την αντίδραση των φορολογουμένων και από την αντίδραση των ε, κυβερνήσεων σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι τελικά η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε χθε είναι πραγματικά καλή συμφωνία. Φυσικά αυτή θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και να, να ζητήσουμε την κατάλληλη νομική βάση. Ποια θα είναι αυτή το άρθρο 122, όπως ανέφερε ο κύριος Ντάφα. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα. Όχι μόνο μιλάει για τις ε, καταστροφές, αλλά και για την ε, αλληλεγγύη. Το άρθρο 136 αφορά την Ευρωζώνη. Και επομένω, οι χώρες που δεν είναι μέλη της ε, Ευρωζώνης δεν καλύπτονται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερα και πιο συγκεκριμένα για την νομική βάση. Ίσως χρειαστούμε και κάποιο επιπλέον άρθρο. Αλλά τώρα πραγματικά κάνω οικοτολογίες. Περιμένουμε τη διμερή διαβούλευση του Προέδρου Φανδρόμπουη με τους εταίρους του. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι επαφές, νομίζω θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για την νομική βάση. Στην Κομισιόν εμείς προτιμάμε μια απλουστευμένη διαδικασία πάντως εν για την ε, έγκριση της αλλαγής της συνθήκης. Θα θυμάστε πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία με την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας και μας ανησυχεί τώρα. Το γεγονός ότι αν χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή αλλαγή, μπορεί να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, μόνο και μόνο επειδή θα κάνουμε κάποιες νέες προτάσεις. Ξανασυζητάμε το, το όλο το πλαίσιο και θα μας, δημιουργήσει μια, θα μας δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Θα ήταν πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία, που είναι πιο στοχοθετημένη. Η αλλαγή θα γίνεται χειρουργικά και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να δίνει νέε εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται, να... Γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ναι. Αν δείτε το μηχανισμό που ξεκίνησε να λειτουργεί για την Ιρλανδία από χθε, ε, βασίζεται και σε διμερεί εγγύησει. Ίσως λοιπόν αυτήν να είναι η λύση. Αλλά και πάλι, η Κάζο εδώ, γιατί ξέρω ότι η ερώτηση του κ. Νταφ ήταν πολύ περίπλοκη. Τώρα για τα δημοψηφίσματα. Αν χρειαστεί να γίνουν δημοψηφίσματα. Είναι θέμα συνταγματική τάξη στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν πώ εγκρίνουν τι αλλαγέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο πάντω είπε ότι αν προκρίνουμε τι απλουστευμένε διαδικασίε για τις αλλαγές ε, των συνθηκών που δεν δίνουν νέε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν υπάρχει και λόγο για δημοψήφισμα. Ήταν μια βρετανική δήλωση πριν από καμιά δυο μέρε. αλλά όλα εξαρτώνται από τη διατύπωση τη πρόταση, ποια είναι η αλλαγή τη συνθήκη που στοχεύουμε και βεβαίω τελικά το λόγο έχουν τα κράτη-μέλη για το πώ θα επικυρώσουν κάτι τέτοιο. Αλλά η προτίμηση της η δική μα είναι η ταχεία, η απλουστευμένη διαδικασία. Γιατί οι λύσει θα είναι, πολύ πιο γρήγορα, θα είναι έτοιμες πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να ξεκινάμε δύσκολες θεσμικές συζητήσεις. Κύριε Τάφα, αναφερθήκατε σε αυτό το σχέδιο, στο νομοσχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μελετάμε. Και θα το συζητήσουμε με τους ε, Βρετανούς ομολόγους μας. Κύριε Μέντες Δεβίγο, για την επικουρικότητα. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, πώς μπορούμε να είμαστε υπόλογοι έναντι των Εθνικών Κοινοβουλίων η επιλογή μας ήταν να ακολουθήσουμε ένα ευρύτερο ε, μια ευρύτερη, μάλλον μια πιο γενναιότερη αν θέλετε προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι ζητούμε απαντήσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια όχι σε ένα νομικίστικο και μόνο και νομικό μηχανισμό αλλά σε, από μια πολιτική ε, πτυχή. Όχι μονάχα να μας λένε αν κάτι εκπληρεί την ε, αρχή της επικουρικότητας ή όχι. Η απάντηση φυσικά βρίσκεται στις νομοδοτήσεις του Εθνικού Κοινοβουλίου. Αν τα Εθνικά Κοινοβούλια θέλουν να σχολιάσουν και το περιεχόμενο του νομοθετήματο, το πρόσφορο ή όχι, την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο νομοθέτημα και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε και όλα τα άλλα ερωτήματα τα οποία θέτουν τα κράτη-μέλη στις ε, ε Απαντήσει στις υποβολέ που μα κάνουν και όχι μονάχα το θέμα του ελέγχου επικουρικότητα. Και οι υπηρεσίε μα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά τα οποία λέγονται στις ε, γνωμοδοτήσει που μα δίνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. πολλέ φορέ είναι πολυσέλιδη η απάντηση και προσπαθούμε να το κάνουμε σαφέ ότι εγώ στέλνω και υπογράφω αυτή την επιστολή, δηλαδή ότι έχει αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή από την Κομισιόν, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις απόψεις των Εθνικών ε, για το προϋπολογισμό του 2011. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αν μπορώ να το πω έτσι, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε, τον προϋπολογισμό, να έχουμε ένα προϋπολογισμό για το 2011 στη διάθεσή μας. Νομίζω όμως ότι όταν υπήρξε η διαφωνία για τον προϋπολογισμό κάποιοι δεν κατάλαβαν τι αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να προκύψουν για τις, παραδείγματος χάρη, τις ε, πληρωμές στους γεωργούς, τις αμέσως πληρωμές οι οποίες προκαταβάλλονται ή την καταβολή πιστώσεων για τα προγράμματα καιροτομίας, έρευνα και ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι υπάρχει από την πλευρά της Κομισιόν μια ισχυρή προτίμηση να υπάρξει μια συμφωνία πριν από το τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο έχει ως εξή. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν εργαστεί πολύ σκληρά και παρουσίασε τη δεύτερη πρόταση του προπολογισμού ήδη την προηγούμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στις 26 Νοεμβρίου. Αναμένουμε τώρα να συζητήσει στις 7 Δεκεμβρίου την πρόταση της Κομισιόν και να την εγκρίνει το Συμβούλιο και ελπίζουμε να υπάρξει ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου, κάτι το οποίο θα κάνει λίγο πιο λαμπερά τα Χριστούγεννά μας και πιο ειρηνικά. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τον προϋπολογισμό στην διάθεσή μας για τις πληρωμές από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και υπάρχουν και κάποιες πληρωμές για την Ισπανία συγκεκριμένα εδώ και επομένως πρέπει να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Μία τελευταία παρατήρηση για την αναλογικότητα στον προϋπολογισμό και την αναλογικότητα στην πολιτική συζήτηση η οποία συνάπτεται με τον προϋπολογισμό. Εγώ πήγα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, είχαμε μια κοινή συνάντηση την επαύριο της αποτυχίας των συζητήσεων των, της για τον προϋπολογισμό και προσπαθούσαν, όπως προσπαθώ όπου και πηγαίνω, όπου να πηγαίνω, ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. 1% από τα οποία 5,7% των οποίων πηγαίνουν για διοικητικές υπηρεσίες, δεν είναι μονάχα οι υπάλληλοι, είναι και οι γλωσσικές υπηρεσίες, είναι οι βάσεις δεδομένων, είναι οι υπηρεσίες τα κτλ. Με 5% το 1% λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή διοίκηση. Είναι μια πολύ καλή προσφορά προς τους Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο του προϋπολογισμού γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις σε εθνικό επίπεδο από τις ε, χώρες μέλη και εμείς θα πρέπει με αλλά με επιμονή να εξηγήσουμε ποια είναι η προστέμενη αξία που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μόνο 1% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρώπης. Πρέπει να το πούμε, να το παραπούμε, να επιχειρηματολογήσουμε και να είμαστε εύγλωτοι για τα θέματα αυτά, γιατί πολλοί στα εθνικά κοινοβούλια αλλά και πολλοί στην κυρία γνώμη της Ευρώπης δεν γνωρίζουν ποια είναι η αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Αποφάσισε η Επιτροπή να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τα, τη πλευρά της διαμάχης περί των προϋπολογισμών Ίνικο και εσύ και άλλος συνάδελφος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα δέκα λεφτά που μας μένουν για αυτό το λόγο. Συμφωνείς. Oh, ναι, ναι, συμφωνώ, λέει ο κύριο Αλλά πρώτα απ' όλα να καθησυχάσω τον κύριο Τιπράτο ότι αυτό που είπα προηγουμένω δεν το είπα για τίποτα έξτρα δαπάνε βάρο τη Κομισιόν τη Ένωση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη σημερινή συγκυρία ορισμένοι εξημών και εννοώ τον φίλων ΝΤΑΦ να συμμετάσχουμε. Και ο κύριος Χριστόφερσον θα πρέπει αυτόν το λάβει υπόψη γιατί τελικά συμφωνήσαμε, είχαμε, έκλεισε το deal, ε, ε, υπήρξε η συνένεση όσον αφορά τον υπολογισμό για πώς το λέμε, πώς το είπαμε, αυτό το πολυετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί πάντοτε εγώ θυμάμαι το, την παλιά ορολογία που έλεγε δημοσιονομικές προοπτικές, οπότε έγινε η διαβούλευση για το κατά πόσον θα έχουμε νέους πόρους, επομένως να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα. Και νομίζω ότι το πιο σωστό θα είναι να προκαταλάβουμε τα πράγματα και να μην θέλουμε να αποσπάσουμε ορθοδιότητες με τρόπο άδικο. Και είναι πολύ σημαντικό να κλείσω ο προπολογισμό και η συμφωνία. Σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει ο φίλο Λεβαντόφσκι να προχωρήσει, όπως είπε. Πώς το είπατε? Πώς το είπατε να, να, να ξεχάσει, να συγχωρήσει, τέλος πάντων. Θα σας πω ότι το ΕΛΚ πάντα χαίρετα σας βλέπει εδώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελε και συνάδελφος να λάβει το λόγο. Αυτό το δεκάλεπτο. Έχετε το λόγο. Τι γίνεται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τι γίνεται με τους φορείς της χρηματοοικονομικής επιτήρησης. Νομίζω ότι το επιβεβαιώνεται πως θα έχουμε προπολογισμό. Και δεν θα πάμε στα 12 τιμόρια. Αλλά με αυτούς τους φορείς τι θα γίνει. Θα δρανίσουμε έχετε κάποια ε, άκρη να μας δώσετε, θα υπάρξει κάποια ε, διέξοδος. Νταφ, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ που απαντήσατε σε αυτό που ερώτησα προηγουμένως. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Για τα θέματα του προϋπολογισμού πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κομισιόν υποστηρίζει την ε, συνέχιση της νομικής ισχύως της διαθεσμικής συμφωνίας του 2006. Ξέρουμε ότι θα αντικατασταθεί εν καιρό με ένα δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά για θέματα όπως το μέσο ευελιξίας έχουμε μια διαθεσμική συμφωνία και πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι ότου αντικατασταθεί από κάτι καινούριο, από κάτι ευρύτερο και πιο μόνιμο. Και σε ό,τι αφορά το πολιετές πλαίσιο δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ε, ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός διάλογος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ινίγκο είχε απόλυτο δίκιο. Ότι εμείς δεν θέλουμε να πετύχουμε περισσότερες εξουσίες πέραν αυτών που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μέσα στην συμφωνία αυτή λοιπόν ήταν σαφές ότι που αποτελεί η Συνδίκη Λισαβόνας, ήταν σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη διατύπωση των πολιετών στόχων και την αναθεώρηση των ιδιών πόρων. Γιατί αν δεν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά πάσαν πιθανότητα Το Κοινοβούλιο με, την... με το τωρινό πνεύμα το οποίο επικρατεί θα απορρίψει και πάλι την ε, θέση του Συμβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Αλλά δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ξέρει ότι θα απορρίψουμε και πάλι μια πρόταση η οποία έχει διατυπωθεί με ένα τέτοιο τρόπο που μας αποκλεί από την πλευρά του Συμβουλίου. Είναι απαραίτητο λοιπόν για την Κομισιόν να αγωνιστεί υπέρ του Κοινοβουλίου στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Yes, thank you very briefly. Πολύ σύντομα. Ως μέλος της Επιτροπής Συνδιαλλαγής για τον Προϋπολογισμό αισθάνομαι την ανάγκη να σχολιάσω και εγώ αυτή την ε, πολύ δύσκολη και μακρά διαπραγμάτευση για τον προπολογισμό που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Καταρχά, συμφωνώ με τον Άντρου Νταφ. Και εγώ θεωρώ παράξενο το γεγονός ότι το, συνομβούλιο, ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι βρίσκεται εκτός της συνθήκης της Λισαβόνας κάτι το οποίο είχε δεχτεί το Συμβούλιο να έχει, δηλαδή, είχε δεχτεί να έχει διαβουλεύσεις. Για άλλα θέματα. Με την επιφύλαξη βέβαια του άρθρου 124 δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα που, συζητάμε, που ζητάμε αυτές τις ε, συζητήσεις ε, από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο μας απαντάει ε, ξεφεύγουν από την συνθήκη. Επίσης, σε αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν, δεν ζητάμε απλώς κάτι παραπάνω. Υπάρχει, να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και το επιβεβαιώνει και η τελευταία πρόταση της Κομισιόν ότι θα χάσουμε ένα εργαλείο που είχαμε μέχρι στιγμής μια ευελιξία. Η, η πρόταση κατεβάζει το κατόφλι. Η πρόταση για την επίλυση των, της κατεπίγουσας ανάγκης. Αν δεν ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτού του κατοφλίου, θα συνεχιστεί η συζήτηση. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε περισσότερες ευθύνες. Λισαβονοποιείται ο προϋπολογισμός και παράλληλα μειώνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε με τη χρήση της ειδική πλειοψηφία αυτή τη μικρή ευελιξία που υπήρχε στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο και παραμένει εκρεμές. Εγώ ομολογώ ότι περίμενα η Κομισιόν να δείξει έτσι πιο να έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα, να είναι πιο επεμβατική κτλ. Μια δύναμη και παθητική κομισιόν δεν είναι καλό για την Ευρώπη. Ε, πρέπει να δείξετε ε, στεναρό πνεύμα, να υπερασπιστείτε την ε, κοινοτική μέθοδο και να παίξετε τον νέο σας ρόλο που σας δίνει η συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μινής. Θα μας δώσετε πέντε λεφτά ακόμα. Δίνω το λόγο στον κύριο Επίτροπο συγγνώμη στον Ινίγκο γιατί σίγουρα δεν ε, εννοούσα αυτό για την ε, Ισπανία. Ήθελα απλώς να δείξω πόσα σχέδια θα φυγούν από την έλλειψη προϋπολογισμού. Εγώ συμφωνώ ότι για το ότι οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ξέρετε πως η ένταση υπήρξε, τη ατμόσφαιρα επικρατούσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά, βρισκόμαστε σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπάθησαμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε μια πρόταση που ελπίζουμε ότι έχει την πιθανότητα να εγκριθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και κάναμε σαφές ότι για τους ίδιους πόρους θα υποβάλει μια πρόταση κομισιόν και θα την υποβάλει μαζί με τις προτάσεις μας για ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του Ιουνίου του 2011. Σε ό,τι αφορά την λισαβονοποίηση του προϋπολογισμού και πάλι ε, μέσα στα πλαίσια της δυσκολίας που υπάρχει καταφέραμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για τα εσωτερικά θέματα και για την ΚΕΠΑ ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και στον τομέα της ευελιξίας, το 0,03 και οι αποφάσεις υπέρ του ITER, πιστεύουμε ότι ήταν το, μεγαλύτερο, το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε σε αυτές τις στιγμές. Υπάρχει φυσικά και η δέσμευση της Κομισιόν να έχει καλύτερη επικοινωνία και καλύτερη επιχειρηματολογία υπέρ της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας η οποία προκύπτει από τον προπολογισμό μα και τη συνεργασία των κρατών μελών. Και επίση θα πρέπει να κάνουμε σαφέ πόσο κοστίζει η μία η μία... μη Ευρώπη, η απουσία τη Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση που έχουμε μπροστά μα. Και εάν τελικά ε, έχει να κάνει με την τήρηση των διαδικασιών, εμεί σεβόμαστε απόλυτα τη συνθήκη και το θεσμικό ρόλο κάθε θεσμικό οργάνο και αυτό περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων μας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τα συγκεκριμένα ερωτήματα τώρα για τις νέες ε, εποπτικές αρχές για, τις, ε, ε, για το πιστωτικό τομέα και εκεί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα προϋπολογισμό. Δεν μπορώ να σας πω ποια, ποιος είναι ο σχεδιασμός μας σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, αλλά σίγουρα θα χρειαζόμασταν να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση για προηγούμενες δομές, για δομές πριν από τη δημιουργία του πλαισίου για την ε, ρύθμιση των αγορών και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για την δομή που υπάρχει τώρα θα ήταν πολύ δύσκολο στην περίπτωση της ΚΑΘΗ να ενσωματώσει τα νέα άτομα από την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων που κανονικά όταν θα ξεκινούσε η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πια. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και αυτή τη στιγμή η νομική υπηρεσία της Κομισιόν ελέγχει τι θα πρέπει να γίνει εάν δεν υπάρχει προϋπολογισμός αλλά ελπίζω ότι θα το αποσύσουμε αυτό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Ζήτα. Και ευχαριστώ και στους που μας βοήθησαν. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνεχίζουμε με την αυριανή συνεδρίαση. Στις 9 το πρωί θα ψηφίσουμε την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο και για την Επιτροπή και για μας. Ευχαριστώ όλη την ε, ομάδα που προετοίμασε το κείμενο. Όσους δεν δω αύριο στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, τους εύχομαι ε, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστή η Πρόεδρος και τους Διερμηνείς. Και εμείς την ευχαριστούμε.